Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Ein gutes neues Jahr wünsche ich allen, weil es die erste Sitzung des Umweltausschusses im Jahr 2010 ist. Herzlich willkommen. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην ε, ακρόαση του ορισμένου Επιτροπού στον τομέα της ε, Περιβαλλοντικής Πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να χαιρετήσω καλύτερα τον κύριο Γιάννη Σποτότσνικ, στην Επιτροπή εδώ. Στις επόμενε τρεις ώρες η Επιτροπή μα θέλει να ε, δημιουργήσει μια εντύπωση κατά πόσον ε, ο υποψήφιο έχει τη δυνατότητα να προωθεί τις εργασία τη Επιτροπή μας, αν έχει μια ευρωπαϊκή σκοπιά και μπορεί να ασχίσει το αξιωμά του άσχετα από οποιοδήποτε συμφέροντα. Επίσης το Κοινοβούλιο θα εκτιμήσει τις ειδικέ γνώσεις του υποψηφίου για το προεπόμενο χαρτοφυλάκιο και την δυνατότητα επικοινωνίας, πράγμα που είναι σημαντικό στην πολιτική γενικά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλος ειδικό. Έτσι αναφέρεται στις κατευθύνσεις γραμμές για τη χορήγηση της σύμφωνης γνώμης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καινούργια Επιτροπή. Ο κύριος Ποτότσνεκ απάντησε γραπτά στις απαντήσεις που του υπήρχε που βάλαμε. Έχετε όλοι, σε όλες τις γλώσσες, τη δέσμη ερωταποκρίσεων στα χέρια σας. Θα ήθελα να σας εξηγήσω την ε, διαδικασία για τις επόμενες τρεις ώρες. Ο υποψήφιος επίτροπος καλείται να κάνει μια δήλωση που δεν επιτρέπει να διαρκέσει πέρα από 10 λεπτά και κατόπιν θα έχουμε 160 λεπτά για ερωτήσεις και απαντήσεις που θα ακολουθούν κάποια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία. Μία ερώτηση. Μία, ένα λεπτό συγγνώμη για την αρχική ε, ερώτηση. Δύο λεπτά για την απάντηση του Επιτρόπου. 45 λεπτά δυνατότητα για συμπληρωματική ερώτηση και ένα λεπτό απάντηση. Μέσα στα πλαίσια αυτών των πέντε λεπτών έχουμε επίσης μια διαδικασία τριών λεπτών όπου προβλέπονται 50 δευτερόλεπτα για την ερώτηση, 2 λεπτά για την απάντηση και καμία συμπληρωματική ερώτηση ή απάντηση προφανώς. Αυτές οι περίοδοι ερωτήσεων τριών λεπτών προβλέπονται στο πρόγραμμα συγκεκριμένα και οι ενδιαφερόμενοι τις γνωρίζουν. Στο τέλος, ο υποψήφιος επίτροπος έχει τη δυνατότητα να κάνει μια δήλωση 5 λεπτών. Εάν κάποιος ε, ερωτών απουσιάζει, διαγράφεται πλήρως η ερώτησή του. Παρακαλώ να είστε παρόντες λοιπόν. Και κάτι άλλο. Η δεύτερη ερώτηση που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρεται στην απάντηση του υποψηφίου επιτρόπου. Δεν επιτρέπεται να αναφέρεται σε ένα δεύτερο θέμα. Ο Προεδρός ε, επιφυλάσσει του δικαιώματο να απορρίψει μια ερώτηση αν δεν ακολουθεί αυτή τη διαδικασία. Και επίση, πολύ σημαντικό για τι επόμενε τρει ώρε, είναι πάρα πολύ στενά τα χρονικά διαστήματα που έχουμε και παρακαλώ τον ε, υποψήφιο επίτροπο να τηρεί και για τις απαντήσεις του το χρόνο αυστηρά, αλλιώς θα αναγκαστώ να παρέμβω με το σφυράκι μου εδώ. Κύριε Ποτόπιν, δεν είσαστε καινούριο στο ευρωπαϊκό, ε, στην ευρωπαϊκή σκηνή. Μέχρι τώρα ήσασταν υπεύθυνο για την ε, έρευνα και αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο και στην πολιτική περιβάλλοντος, τεχνολογία παραδείγματο χάρη ή τεχνολογία καθαρών καυσίμων, που όλα αυτά υπάρχουν νέα ερωτηματικά για τον νέο επίτροπο. Και ακριβώς τώρα στις αρχές του 2010, όπου ο κύριος Παρόζο έχει χωρίσει τα φαρτοφυλάκια ένα για τις κλιματολογικές αλλαγές και ένα για την ενεργειακή πολιτική, είναι πάρα πολύ σημαντικό η ευρωπαϊκή ε, πολιτική περιβάλλοντος να έχει ένα δικό της προφίλ, να είναι ανεξάρτητη, να έχει ένα δικό της όραμα. Περιμένουμε να ακούσουμε με ενδιαφέρον τις ιδέες σας για την περιβαλλοντική πολιτική κατά διάρκεια της δίας Έχει το λόγο κύριε Ποτότσνικ. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί βουλευτές, είναι σπάνια ευκαιρία ε, για μένα διότι συνήθως σλοβενικά δεν μπορώ να μιλήσω στους διαδρόμους της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής οπότε θα σας μιλήσω στην ε, γλώσσα μου και όμως μετά πρόκειται να σας απαντήσω ρωτή σας ή στα αγγλικά. Κύριε Πρόεδρε Λάινεν, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, το σωστό για κάποιο υποψήφιο, για κάποια δημοσία θέση μεγάλες ευθύνες είναι τον εμφανίζεται κάποιου συνοποιών σα και αυτόν τον τρόπο εσά που είσαστε οι άμεσα εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Ευρωπαίων Πολιτών. Και επίση θα πρέπει να απαντήσω στι ερωτήσει σα. Γνωρίζω επίση ότι αν ο ορισμό μου επικυρωθεί ή κυρωθεί, όχι μόνο θα έχω την εμπιστοσύνη σα, αλλά θα έχω και αξιοπιστία εναντί του κοινού, εναντί του κόσμου. σω κάποιοι από εσά με γνωρίζουν και έχουμε συναντηθεί με ορισμένου από εσά που έχουμε τη Σλοβενία την τελευταία πενταετία. Διετέλεσα επίτροπο για τα θέματα επιστήμης και έρευνα Εσεί γνωρίζετε ότι έχω ε, σπουδάσει οικονομικά και ήμουν επικεφαλή των διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ το βόλιο Και έχω και δύο παιδιά, δύο γιους. Και ξεκινώ με ε, την εξή ρίση γνωμικό ότι η Ευρώπη είναι μια μεγάλη ήπειρος και ή θα είναι μεγάλη ήπειρος ή δεν θα είναι τίποτα. Και το ίδιο ισχύει και για το σύνολο της υδρογείου. Ε, όσον αφορά την οικολογία των, των λεγόμενων μπλε γαλάζιο πλανήτη. Ή θα είναι γαλάζιος ή τίποτα. Και οπότε θα σα παραπέμω σε όσοι το 2008, γιατί τότε ω επίτροπο για το χαρτοφυλάκιο που σα είπα, ε, είχα εμφανιστεί βιών σα και με είχατε τότε εγκρίνει. Οπότε ε, θα πρέπει να σα πω ότι το θέμα τώρα η λέξη κλειδί είναι η βιωσιμότητα με κάθε έννοια του όρου. Κάτι το οποίο αφορά το περιβάλλον, αλλά επίση σημαίνει πάρα πολλά για τον κόσμο που τον καίει, του Ευρωπαίου πολίτε και η Ευρώπη. Δεν είναι κάτι το οποίο βγαίνει από μια συνθήκη, από ένα εγχειρίδιο είναι κάτι το οποίο αφορά την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων σε πόλεις, σε περιφέρειες και σε χώρες και οι κανόνες και οι νόμοι της Ευρώπης ε, λειτουργούν ε, για τους ε, Ευρωπαίους οπότε και έτσι αποκτά κάποιο πλεονέκτημα, κάποιο ατού η Ευρώπη που πριν από λίγες δεκαετίες βρισκόταν σε ερήπια, χρειαζόταν κάποιο είδους ανασυγκρότηση και ήταν απελπισμένος ο κόσμος, χρειαζόταν την συμφιλίωση οπότε η ε, συνεργασία ήταν κάτι το αυτονόητο και παράμα αυτονόητο. Και έφερε ειρήνη και ασφάλεια η ΕΕ. Και ε, τέτοια κίνητρα ε, ήταν πίσω από τι πράξεις των προκατόχων μα πριν από μια πεντηκονταετία. Όμω, σήμερα τα βλέπουν αλλιώ οι νέοι. Λένε ότι στην Ευρώπη τα περνάμε ωραία γιατί τότε να γίνει πιο στενή η συνεργασία μα. Όχι, πρέπει να γίνει πιο στενή διότι δεν έχει αλλάξει μόνο η Ευρώπη. Έχει αλλάξει όλο ο κόσμο και άλλαξε με τρόπο εντυπωσιακό, δραματικό και έχει αλλάξει χωρί ε, επιστροφή. Είτε μα αρέσει είτε όχι, όλο ένα και μεγαλύτερη είναι η αλληλεξάρτηση. Και ε, βεβαίως απολαμβάνουμε τα θετικά της παγκοσμιοποίηση, αλλά υφιστάμεθα και τα προβλήματα αλλαγή του κλίματος, τα προβλήματα τα ενεργειακά, τι επιδημίε, το, το ότι δεν έχουμε βιοπικιλότητα πια, ε, ελλείψεις σε, σε, σε είδη διατροφής, νερό, τις διορθωτικές οικονομικές ανισορροπίες, την ανασφάλεια. Όλα αυτά επομένως είναι προβλήματα κοινά. Είναι προβλήματα που αφορούν όλους και αυτές οι νέες προκλήσεις έχουν ανεβάσει τον πύχη όσον αφορά την κοινή υπευθυνότητα και την ατομική υπευθυνότητα. Οπότε αυτό που θα πρέπει να πούμε στους Ευρωπαίους για αυτές τις προκλήσεις είναι το ότι θα πρέπει να έχουμε μια προσπάθεια αποδοτική μόνο εάν κινηθούμε από κοινού. Και ο πρώτος, 21ος αιώνας είναι ο αιώνας του, του, εφήμερου και θα πρέπει όμως το εφήμερο το κάνουμε βιώσιμο και γι' αυτό να έχουμε μια παγκόσμια διακυβέρνηση οπότε θα χρειάζεται μια υπεύθυνη Ευρώπη, μια Ευρώπη που μπορεί να έχει μια φωνή και που μπορεί να, να κρατήσει τα, τα ενία της ε, πολιτικής πρωτοπορίας και θεωρώ ότι ε, εγώ πρεσβεύω μια τέτοια Ευρώπη και νομίζω ότι με τέτοια πρέπει να ταυτιστούν οι νεότερε γενιέ. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα, στο, στη μέση μια διαδρομή μετασχηματισμού μετά τον πόλεμο, μετά από μια οικονομία που ξεκίνησε η οικονομία των φυσικών και άλλων πόρων και, ξεκίνησε, και κατέληξε η οικονομία τη γνώση και το ξεκαθάρισε ο πρόεδρο Μπαρόσο ότι ε, να ταινίζουμε την ΕΕ του 2020, αλλά χρειάζεται μια προσέγγιση πιο πολύ, πιο πολύ σύγκληση και οπότε θα πρέπει να δούμε ποια είναι η ειδική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ, εγώ λέγω, πρεσβεύω αυτούς τους στόχους και πιστεύω ότι με τη συνθήκη της Λισαβόνας θα έχουμε μια εταιρική σχέση που είναι πιο σημαντική περισσότερο από ποτέ. Και σας μίλησα για έναν ευάλωτο κόσμο και ακριβώς αυτή η ιδιότητα του, του ευάλωτου κάνει το περιβάλλον κάτι το οποίο είναι θέμα κλειδί για το μέλλον. Τι είναι πιο σημαντικό, τι είναι πιο παγκόσμιο ε, από το ότι θα πρέπει να φροντίσουμε τον αέρα που αναπνέουμε, τη γη στην οποία πατάμε και το νερό που πίνουμε. Γιατί κάποια εποχή μίλαγε ο κόσμο για βιώσιμη ανάπτυξη και μίλαγε για το περιβάλλον σαν ένα θέμα διοντολογικό, ηθικό και κάτι το οποίο απασχολούσε κάποιους σπεσιαλίστε, κάποιους περιθωριακούς, Τώρα όμως τα πράγματα δεν ισχύουν αυτά. Τώρα θεωρούμε ότι ο οργανισμός για το περιβάλλον είναι κάτι το οποίο καίει όλο το πολιτικό φάσμα. Τώρα θα πρέπει να πείσουμε ε, τον κόσμο για το ότι υπάρχουν πιστικές ε, ε, ενδείξεις ότι εμείς ίδιοι έχουμε καταστρέψει το περιβάλλον. Οπότε η ολόκληρη γενιά Ευρωπαίων τώρα ζητεί ξεκάθαρη ανάληψη δράσης και θα πρέπει να αναστρέψουμε ναι. αυτήν την και να την αυτή την καταστροφή που επιφέραμε στον πλανήτη μα. Δεν είναι λοιπόν κάτι το οποίο αφορά τι μέλου γενία είναι κάτι που αφορά τη δική μα γενιά. Και επίση ε, υπάρχει και αυτό το θέμα του ότι η προστασία του περιβάλλοντο φέρνει και κάποια ωφέλη οικονομικά, κοινωνικά, επιχειρηματικά δεν ε, θα βγούμε άλλο τρόπο από την, από την κρίση. Δεν μπορώ να, φυσικά να αρνηθώ. Ο υποστήριο περιβάλλοντο ε, κοστίζει. Ε, είναι θέματα νομοθετικά, είναι θέματα διοικητικά. Όμω μακροπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα φέρνει εξοικονόμηση δαπανών. Επίση βελτιώνει την ποιότητα τη ζωή, τονώνει την οικονομία και δημιουργεί θέσει εργασία. Φυσικά και χρειαζόμαστε νέε θέσει εργασία. Άλλοι χρειαζόμαστε ανάπτυξη, χρειαζόμαστε συνοχή, βιώσιμη ανάπτυξη, χρειαζόμαστε μία οικονομία που αποδεύεται αποτελεσματικά τους πόρους και βασίζεται στη γνώση. Εγώ, ως Επίτροπος Περιβάλλοντος, θέλω αποτελέσματα. Και τι εννοώ. Οι Ιαπωνέζοι λένε ότι το όραμα χωρίς πράξη είναι σαν κανένας να ονειρεύεται. Και χρειαζόμαστε επομένως μια ένα τέτοιο όραμα, χρειαζόμαστε πολιτικές, ε, που θα στηρίζονται σε στοιχεία ατράνταχτα. Επίση θα πρέπει να ποιε είναι οι καλύτερε πολιτικέ, τα καλύτερα εργαλεία για αυτέ τι πολιτικέ που και αυτέ θα βασίζονται σε στοιχεία ατράνταχτα. Διότι το περιβάλλον είναι κάτι περίπλοκο όπω και ο ίδιο ο κόσμο. Και ακριβώ γι' αυτό το λόγο όλα αυτά τα θέματα του περιβάλλοντο επικαλύπτονται με άλλε ευθύνε και άλλου είδου συμφέροντα και ενδιαφέροντα. Γι' αυτό, εάν εγώ πρόκειται να πετύχω κάτι συγκεκριμένο σαν επίτροπο για το περιβάλλον, αυτό ε, δεν θα, θα γίνει μόνο εάν κάνω κάτι για να διατηρήσω απλώς τα, τα, τα κεκτημένα σε αυτό το χώρο. Οπότε και εγώ θα δώσω μια μάχη σκληρή, ούτως ώστε να έχουμε προσέγγιση ε, συνεκτική, λογική, συνεπή για όλες τις πολιτικές και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα οικονομικά μέσα που έχουμε στην ε, διάθεσή μας για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους και γι' αυτό θέλω να έχουμε καινούργιες συνεργασίες με τα κράτη-μέλη, με άλλες περιφέρειες, η επικουρικότητα να μην είναι μια, μια, μια πρόφαση, μια δικαιολογία αδράνειας όμως θέλω από κοινό να πετύχουμε για ποιου στόχου και γι' αυτό και θέλω να συνεργαστώ με όλου εκείνου οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν τόσο ώστε να βελτιωθεί η υπόθεση περιβάλλον και ο διάλογο να είναι ένα όπλο, ένα όπλο αποτελεσματικό. Διάλογο και με εσά, αγαπητοί βουλευτέ. Με μη κυβερνικέ οργανώσει, με τι επιχειρήσει, με του Ευρωπαίου και με του διεθνεί μα εταίρου. Θέλω πολιτική για το περιβάλλον να ε, είναι όσο γίνεται πιο τεκμηριωμένη ε, και να περνάει μέσα από ένα αποτελεσματικό διάλογο. Θέλω να υπάρχει αποτελεσματικότητα, να υπάρχει συνένεση, να, είναι, να υπάρχει το, το mainstream σε όλες τις πολιτικές, αλλά να είναι πρακτική και να είναι στοχευμένη. Τώρα να σας πω τους βασικούς άξονες της μέλους σας δράσης μου. Πρώτα-πρώτα αποτελεσματικότητα. Η προτεραιότητά μου θα είναι να εξασφαλίσω ότι το, το όραμα για την ΕΕ του 2020 θα κατατείνει στο να έχουμε ανάπτυξη, να έχουμε θέσεις επασχόλησης, να έχουμε γερά θεμέλια, να έχουμε βιωσιμότητα και αποτελεσματική χρήση των πόρων. Να επικεντρωθούμε όσον αφορά τη σχέση μεταξύ ανάπτυξη και χρήση των πόρων, κάτι το οποίο πρόκειται να αναφέρει αλλαγή της συμπεριφοράς μας και στην κοινωνία και στην οικονομία, κάτι το οποίο είναι δύσκολο αλλά εφικτό. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι ε, ήδη είναι εφικτό γιατί ήδη για τι επιχειρήσει η αποτελεσματικότητα είναι η δεύτερη φύση. Αλλά θα πρέπει να, να δούμε πώ αυτή η έννοια θα γίνει πιο ελκυστική θα πρέπει όμως να έχουμε μια πράσινη οικονομία, θα δώσουμε σκληρή μάχη, να βρούμε τρόπου ώστε να αξιοποιήσουμε το περιβάλλον και να το λαμβάνει υπόψη στην λήψη αποφάσεων. Θα πρέπει να δούμε ε, το, το, το, ότι η επιβίωση όλων των ειδών στη φύση είναι κάτι το οποίο μας κάνει πιο πλούσιους για μας και το, για το περιβάλλον. Άρα θα θέλουν τέτοια νομοθεσία ε, και νομοθεσία που να φέρνει καλύτερη ποιότητα ζωή και περισσότερη ευημερία. Δεύτερο άξονα για τη δράση μου θα είναι η βιοπικιλότητα. Κάτι το οποίο χρειάζεται, ώστε να μπορέσουμε να την ε, βοηθήσουμε, να κάνουμε κάτι για να ανασχέσουμε την ε, υπερβολική θέρμανση του πλανήτη, την αλλαγή του κλίματος και πιστεύω ότι τώρα που έχουμε διαφορετικά χαρτοφυλάκια που ασχολούνται με το, με το, με το κλίμα, με την, με την οικολογία, θα μπορούσαμε να πετύχουμε περισσότερα. Τρίτον, τρίτο άξονα είναι η εφαρμογή, η εκτέλεση της νομοθεσίας, η είδη. Ε, πρέπει να δούμε ότι πετυχαίνουμε πολλά εάν φροντίσουμε τα, το, το, το, κείμενο νομοθεσία να εφαρμόζεται, αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο το γράμμα του νόμου, θα πρέπει να υπάρχει ε, ασφάλεια δικαίου, θα πρέπει να υπάρχει προβλεψιμότητα, γιατί αυτά χρειάζεται ο επιχειρηματικός κόσμος, αυτά προσδοκά από εμάς. Έχετε και ξεπεράσει τον ε, χρόνο σα, δεν θα προφτάσουμε. Τώρα θα προχωρήσουμε και θα απαντήσετε στι ερωτήσει. Εάν δεν χρησιμοποιείτε πολύ ε, πολύ λυγική γλώσσα, θα μπορούσαμε να τηρήσετε ένα λεπτό. Ελπίζω όπως και το, στο βόλιο να περάσετε την μπάλα γλίγορα. Κρυσέφερ του ΕΛΚ ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε, κύριε Επιτροφέ, κύριε υποψήφια Επιτροφέ. Έχετε το δυνατότητα να αναφέρεστε σε αυτά που ήδη είχατε πει ήδη στο παρελθόν. Και επίσης ξέρετε πολύ καλά τη διαδικασία της ακρόασης. Κάτι έχει αλλάξει όμως, γιατί στο παρελθόν ε, λέγαμε ότι θα πρέπει να είναι κανένας οδυνατόν μη ακριβής και θα ικανοποιείται το Κοινοβουλίο. Τώρα όμως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εμείς είμαστε όλοι υπέρ της έρευνα και της ανάπτυξης. Είμαστε όλοι υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν όμως διαφορές μεταξύ και των θεσμικών οργανών και των πολιτικών ομάδων. Και αν αναφερθώ σε κάτι που είπατε στη γραπτή σας απάντηση και σε αυτό που είπατε τώρα. Ε, βλέπω ότι πολλά καλύπτεται, αλλά σας παρακαλώ στην ακρόαση αυτή να μας δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις. Ιδίω όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την πολιτική για τους πόρους. Ένας πολύ κεντρικό τομέα, αυτό που με ενδιαφέρει ιδίω εδώ, είναι ο τομέας του ύδατος. Να μας πείτε ότι θα υπάρχει κάποια στιγμή κάποια πρόταση, δεν αρκεί. Ο κύριος Πατώσχη. Uh, Νομίζω πως είναι ένα από τα πράγματα που έμαθα ενώ μελετούσα κατά τη διάρκεια που ήμουν ελεύθερος ότι δηλαδή η προσέγγιση προς τα περιβαλλοντικά θέματα θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε οριζόντια. Και είμαι βέβαιος ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα με ολιστικό τρόπο. Πολλά πράγματα που είναι απαγορευτικά, είναι, είναι μάλλον ε, μέτρα απαγορευτικά, εξαρτώνται από, μα... από μένα, ενώ τα κίνητρα εξαρτώνται από συναδέλφους. Ε, θα πρέπει λοιπόν να γίνει συνδυασμένη προσέγγιση. Ε, όταν δούμε τώρα την νομοθεσία που έχουμε για τα ύδατα και γενικά για το περιβάλλον, πρόκειται για 250 νομοθετήματα. Το νερό και τα απόβλητα είναι τα πιο περίπλοκα, αλλά πιστεύω πως έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα και θα μπορέσουμε να πετύχουμε και αρκετά για το μέλλον. Αυτό που θα ήθελα να, κάνουμε για το, να κάνω άμεσα για το νερό είναι να δούμε σε πόσο έχουμε προχωρήσει τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2012 να έχουμε έναν χάρτη για την ε, διασφάλιση και την προστασία των ευρωπαϊκών υδάτων, ώστε να έχουμε μία προσέγγιση βασισμένη συμβαίνει στις ε, λεκάνες των ποταμών, πράγμα το οποίο εισάγεται μέσω της νέα ε, νομοθεσίας περί υδάτων, ε, να ασχοληθούμε περισσότερο με την εξοικονόμηση υδατος, να εστιάσουμε την προσοχή στην διαθέσιμότητα του νερού και την αντίσταση στο κλίμα. Νομίζω πως αυτό δεν θα γίνει μεγάλη κλίμακα ανανέωση της ε, νομοθεσίας περί ύδατος. Θα διακόπτει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. και. Συμπληρωματική ερώτηση, ο κύριος Ζήβερ, μάλλον πρώτα. Αν κατάλαβα καλά κύριε Επίτροπε. Εσεί είσαστε ικανοποιημένοι με την επανεξέταση τη οδηγίας για τα ύδατα. Δεν θέλετε να κάνετε τίποτα άλλο. Δεν θα ασχοληθείτε καθόλου με πλημμύρε, παραδείγματο χάνει και τέτοια που οφείλονται στι κλιματολογικέ αλλαγέ. Άρα μην ξεχνάμε, η βιομηχανία χρειάζεται νερό, η γεωργία χρειάζεται πορό. Υπάρχουν πολλέ περιοχέ που βρίσκονται σε στρε όσον αφορά το είδωρ πραγματικά είναι ικανοποιητική η εφαρμογή τη οδηγία για το είδο και δεν χρειάζονται συμπληρωματικά μέτρα και άλλη ερώτηση συμπληρωματική. Στην επόμενη χρηματοδοτική περίοδο θα προβλέψετε περισσότερου πόρου, οικονομικού πόρου στον τομέα του του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. We don't have only water framework directive. We have uh, Δεν έχουμε μόνο ε, την ε, οδηγία για τα είδατα, έχουμε και για τα απόβλητα και για τα ύδατα ε, των ε, αστικών περιοχών κλπ. που υπάρχουν προβλήματα. Ε, Παραδείγματος για τα ε, απόβλητα και τα λύματα στις αστικές περιπτώσεις. Μετά έχουμε την οδηγία για το θαλάσσιο πλαίσιο. Πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά στο μέλλον. Δεν νομίζω ότι έχουμε επιλύσει τα πάντα. Όχι. Αλλά θα ήθελα να εξετάσουμε το θέμα αυτό με σωστό οριζόντιο τρόπο. το ερώτημα που θέσετε για την οικονομική ε, υποστήριξη είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά θα πρέπει να φταστούν πολλά από τα θέματα. Ε, η γεωργική πολιτική, η κοινή γεωργική πολιτική, είναι μετά στις διαθωτικές ε, πολιτικές κλπ. Είναι πάρα πολύ σημαντική λοιπόν η συνεργασία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τώρα Ελίνα Μακέβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλώς ορίσατε κύριε υποψήφι. Ξέρετε πως ε, το σημαντικότερο είναι όχι μόνο τα λόγια εδώ μέσα ε, στο Κοινοβούλιο, αλλά είναι σημαντικότερα ακόμα περισσότερο για, τους, για το κοινό, για τους ψηφοφόρους μας. Και πολλές από τις ερωτήσεις που έχουμε εδώ συντάξει βασίζονται στις δικές τους ερωτήσεις. Μιλήσατε για το δικό σας όραμα και είπατε ότι δεν θα σπαταλήσετε χρόνο και θα αντιμετωπίσετε τα βασικότερα περιβαλλοντικά θέματα. Ποιο πιστεύετε πως θα είναι το κληροδότημά σα μετά από πέντε χρόνια ως περιβάλλον, περιβάλλοντο. Περιβάλλοντος. Ο κύριος Δήμας αφήνει ένα σοβαρό κληροδότημα όσον αφορά την νομοθεσία περί κλιματικών αλλαγών. Εσείς τι θα θέλατε να αφήσετε πίσω σας. Υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία είναι ε, συνεπή, δηλαδή δύο, λεπτά έχω μόνο, ενώ η ερώτησή σας είναι πολύ ευρία. Εγώ πιστεύω ότι ένα από τα θέματα τα οποία θέλω να υπογραμμίσω και που συνδέεται επίση με την ζωή μου ως επίτροπο σε αυτή την επιτροπή είναι καταρχήν ήθελα θέλω να αυξηθεί η πολιτική προσοχή και η πολιτική υποστήριξη καθώς και η κατανόηση για τα θέματα αυτά. Επίσης η, ενημέρωση του κοινού είναι πολύ σημαντικό. Όλα αυτά τα θέματα που υπογράμμισε ως προτεραιότητες είναι πολύ σημαντικό να κατανοηθούν και από το, από το κοινό. Και ένα από τα θέματα που ήταν πιο δύσκολα είναι ότι εξετάσαμε τα θέματα της έρευνα και της ανάπτυξης περισσότερο από την προοπτική της ε, τωρινής της αγοράς οικονομίας. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όταν διαχειριζόμαστε θέματα ανάπτυξης και απασχόλησης θα πρέπει χέρι με χέρι να τα εξετάζουμε μαζί με τα θέματα έρευνας και ανάπτυξης και το ίδιο πρέπει να συμβεί και με το περιβάλλον και νομίζω πως είμαι σε θέση να το πράξω αυτό. See, you have one more minute. Θέλω να ζητήσω από τις υπηρεσίες να βάλουν στην άκρη λίγο το, την οθόνη για να μπορεί να βλέπει και ο υποψήφιος επίτροπος την ώρα που περνά. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικά θέματα όπου μπορώ να δώσω προστιθέμενη αξία. Δηλαδή να συνδυαστεί, να υπάρχει μια γενικότερη και ολιστική προσέγγιση Πιστεύω ότι υπάρχει χώρος για ελιγμούς. Δεν ε, είμαι άνθρωπος που θα προσπαθήσει να σας δώσει κάτι σε μισό χρόνο ή σε ένα χρόνο. Είναι σημαντικό βέβαια να γίνουν βήματα γρήγορα για τα θέματα που είναι επιτάπητος, αλλά αυτό που μετρά είναι η απογραφή που θα γίνει στα πέντε χρόνια και σε αυτά τα πέντε χρόνια θα ήθελα να θυμάστε αυτή την περίοδο ως μια περίοδο όπου πραγματικά θα έχουμε κάνει καλή δουλειά για το περιβάλλον. Εντάξει, ο Κρις Ντέιβις. όχι, συμπληρωματική ερώτηση. Ναι, πρέπει να το συνηθίσω, με συγχωρείτε. Αναφέρατε την απασχόληση, γιατί βέβαια αυτό είναι προτεραιότητα με την οικονομική κρίση για όλους μας. Πώς απαντάτε σε εκείνους που λένε ότι δεν, μπορούμε να επενδύσουμε στο περιβάλλον αυτή τη στιγμή γιατί προηγούνται οι θέσεις απασχόλησης. Μα επενδύοντας στο περιβάλλον ε, βάζουμε πρώτες τις θέσεις απασχόλησης. Αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο για όλους. Ο καλύτερος τρόπος για να το εξηγήσουμε είναι μέσω της ε, ιστορίας για τις κλιματικές αλλαγές. Το πραγματικό ζήτημα όταν κανείς για να, ασχολεί, για να αντιμετωπίσει αυτά τα πράγματα είναι να καταλάβει πως η κλιματική αλλαγή είναι πλέον πραγματικότητα. Αν η απάντησή μας σε αυτή την ερώτηση είναι ναι, οι κλιματικές αλλαγές είναι πραγματικότητα και προκαλούνται από τους ανθρώπους, ε, τότε βεβαίω οι απαντήσει που συνδέονται με το πώ θα πρέπει να αντιδράσει ο επιχειρηματικό κόσμο είναι ξεκάθαρε. Όποιο πρώτο ασχοληθεί με αυτή τη δουλειά θα είναι και αυτό που θα κερδίσει. Και η δική μας ε, ε, δουλειά είναι να δώσουμε σαφή μηνύματα ότι αυτό αυτή είναι η κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε. Δεν χρειάζεται να είμαστε ευγενικοί. Χρειάζεται να είμαστε προβλε... θέλουν να έχουν στη διάθεσή τους προβλέψιμες και μακροπρόθεσμες θέσεις. Αν το καταφέρουμε αυτό θα με κάνει σωστά τη δουλειά μας. Ευχαριστώ. Ο Κρίς Davis. Κύριε Πίτροπε, τι εναρκτήριέ σα ομιλίε μπορεί να μην κρατήσατε το χρόνο, αλλά μου αρέσαν τα λόγια που χρησιμοποιήσατε και είχα την εντύπωση πω ήταν από καρδιά. Μπορείτε να μας ονομα... να κατονομάσετε οποιοδήποτε άτομο σε ολόκληρο τον κόσμο που να έχει δυναμικό για να προωθήσει ε, τις καλές πρακτικές για το περιβάλλον όσο δύναμη έχει ο Επίτροπος για το περιβάλλον της Κομισιόν. Ε, το ρωτώ αυτό για να δω αν έχετε, υπόψη, αν έχετε πραγματικά συνειδητοποιήσει πόσο σημαντική είναι η θέση σας για ολόκληρο τον υδρόγειο. Δηλαδή, τι θα κάνετε, θα γίνετε ακόμα ένας επίτροπος που θα ε, προωθεί οδηγίες στο σύστημα ή θα παίξετε ηγετικό ρόλο και θα υποστηρίξετε σε ολόκληρο τον κόσμο τις ε, βιώσιμες πρακτικές για το περιβάλλον που εσείς υποστηρίζετε. Η σύντομη μου απάντηση είναι ναι, αλλά επειδή έχω δύο λεπτά ε, αναπτύξω περισσότερο την απάντηση αυτή. Είμαι βέβαιος ότι αργότερα θα με ρωτήσετε αργότερα γιατί το χαρτοφυλάκιο για το περιβάλλον ήταν ένα προηγουμένως ενώ τώρα είναι δύο που έχει χωριστεί στις κλιματικές αλλαγές και το περιβάλλον. Αλλά πραγματικά όταν ε, μελέτησα όλα όσα συνδέονται με το περιβάλλον πιστεύω πως είναι τόσο πολλά που το να έχει κανείς ξεκάθαρη εικόνα ε, σχετίζεται με το θαύμα. Όταν ρώτησα τον προκάτοχό μου τον Επίτροπο Δήμα. Πόσο δουλειά είχε με το περιβάλλον, η απάντηση ήταν όσοι ακριβώς θέλεις έχεις». Πάντα υπάρχει δουλειά. Ε, ξέρω πολύ καλά ότι είμαι σε θέση να είμαι ανάμεσα στους ηγέτες του κόσμου, αλλά πρέπει να προειδοποιήσω ότι δεν είμαστε οι μόνοι οι οποίοι κατανοούμε, που κατανοούμε ότι ο κόσμος αλλάζει. Υπάρχουν πολύ σημαντικές αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στην αντιμετώπιση αυτού του έφραυστου, όπως σας είπα, κόσμου. Ε, ίσως ορισμένοι άλλοι να μην το κάνουν με τον ίδιο ακριβώ τρόπο. Ίσως να εστιάζουν ας πούμε περισσότερο σε άλλα στοιχεία, τεχνολογική ανάπτυξη ας πούμε αντί τη συμπεριφορά μας. Εγώ πιστεύω πως και τα δύο χρειάζονται. Πιστεύω πως μια ταυτόχρονη προσέγγιση είναι πολύ σημαντική. Αλλά δεν πρέπει επίση να υποτιμάμε ότι και άλλοι υπάρχουν που καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Θα πρέπει να προωθήσουμε τη δική μα ατζέντα και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μείνουμε σε ηγετικό ρόλο. Αν όμως κάτι σαν την Κοπεχάγη συμβεί, δεν θα πρέπει να θα, θα, πρέπει να επανεξετάσουμε τα σχέδιά μας και τις δεσμεύσεις μας, θα πρέπει να τα θέσουμε επιτράπητος και θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να κάνουμε και τους υπόλοιπους να συμφωνήσουν. Και από αυτή την άποψη, όντως ο ρόλος μου στον τομέα του περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντικός. Ναι. Επερώτηση. Μην ανησυχείτε, δυόμιση ώρες έχουμε ακόμα. Λοιπόν, Έχουμε όμως, ε, πρέπει να, να, να, να θέτουμε σε εφαρμογή τα όσα διακηρύσουμε. Έχουμε πολλά που δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη όσον αφορά την ε, περιβαλλοντική νομοθεσία. Οι διαδικασίες επιβολής της Κομισιόν δεν, είναι πολύ, δεν δίνουν πολλά κίνητρα, είναι εξαιρετικά νομικίστικες Και ε, η Κομισιόν μέχρι στιγμής δεν έχει καταδείξει τις, την αποτυχία των κρατών μελών, δεν, τα, δεν έχει προωθήσει. Ε, θα πιέσετε ώστε να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Είστε έτοιμος να, να κατονομάσετε αυτούς που δεν καταφέρνουν να επιβάλλουν την περιβαλλοντική νομοθεσία. Κοιτάξτε, η προσέγγιση μου ως προς αυτό θα ήταν ε, διφύς. Δηλαδή, εάν έχουμε υιοθετήσει νομοθεσία, οφείλουμε να την ε, ε, εφαρμόσουμε. Δεν υπάρχει ζήτημα. Στο κάτω-κάτω όλοι την έχουμε συμφωνήσει. Εμείς και τα κράτη... Εσείς μάλλον, το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη και έχουν δεσμευθεί ε, νομικός μου λοιπόν ο ρόλος είναι να την επιβάλλω και αυτό σκοπεύω και να κάνω. Από την άλλη πλευρά είναι φυσικά εξαιρετικά σημαντικό να προσφέρουμε και μια χείρα βοηθεία στα κρατημέλη όταν αυτό είναι δυνατόν όταν δεν υπάρχει ε, επαρκής κατανόηση, όταν μπορούμε να μοιραστούμε τη γνώση και τα καλά μας παραδείγματα. Αυτό πρέπει να το κάνουμε. Με ερωτήσαν ε, σε μια συνέντευξη στη Σλοβανία για το περιβάλλον. Βεβαίω η απάντηση ήταν ότι δεν μπορώ να απαντήσω αυτή τη στιγμή γιατί δεν έχω ακόμα εκλεγεί. Αλλά, βάση περιπτώσει, η ερώτηση ήταν αν και, και πώ μάλλον θα αντιδρούσα αν έπρεπε να ενεργήσω κατά τη Σλοβενία. Η απάντησή μου θα ήταν πολύ απλή. Θα ενεργούσα όπω και έναντι από οποιοδήποτε άλλο κρατό. Γιατί, επειδή είναι προ το συμφέρον όλων των πολιτών και των Σλοβαίνων συμπεριβαλλονμένων. Παρακαλώ να μένετε στο ένα λεπτό για να μην χάνουμε περισσότερο χρόνο. Jag ställer på svenska. Swedish. Vi tar ett specifikt... Στα σουηδικά. Εδώ υπάρχει ένα ξεκάθαρο παράδειγμα, δηλαδή η εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικής με το ΡΙΤΣΑ. Είναι πάρα πολύ ε, βασική προσπάθεια αυτή, ούτως ώστε να μην έχουμε κάποιες βλα, βλαβερές ουσίες στην ε, ατμόσφαιρα, ε, στο περιβάλλον γενικότερα. Όμως, κατέληξε αυτή η ιστορία σε κάποιο σκάνδαλο. Εσείς τι θα κάνετε, τι λέτε. Έχουμε πρόβλημα επίσης και με τους ορισμούς που περιέχονται στα παραρτήματα της νομοθεσίας της σχετικής με το ΡΙΤΣ. Όμως, έχουμε τη σύμβαση POPS, τη συνθήκη POPS της Στοκχόλμης. Πρόκειται να κάνετε αναθεώρηση της της εν λόγω συνθήκης για τους ορισμούς των σχετικών βλαβερών ουσιών. Πρώτα πρώτα να σας πω αυτό το οποίο πιστεύω καταρχήν σαν την δέουσα προσέγγιση της νομοθεσίας που έχουμε θεσπίσει. Η εφαρμογή νομοθεσία δεν πάει να πει νέες διαπραγματεύσεις σε σχέση με το πώς θα πρέπει να είναι η η, η, η νέα συνθήκη. Γίνανε τέτοιες ε, ε και άρα θα πρέπει τώρα να ενεργήσουμε εις το πνεύμα και το γράμμα και των διαπραγματεύσεων. Έχουμε που είπαμε εδώ πέρα 50 τέτοιες σχετικές ουσίες, 7 εξ αυτών ε, είναι στην πρώτη δέσμη Καμία δεν είναι στο, στο παράδειγμα 14, οπότε δεν έχουμε εδώ κανένα πρόβλημα. Λέω όμως Ήδη έχω απευθυνθεί εις τον κύριο Ταγιάννη, τον συνάδελφο που έχει το σχετικό το χαρτοφυλάκιο και θα συνεργαστούμε, θα προσπαθήσουμε να τα πετύχουμε όλα όσα θέλουμε, γιατί πρόκειται για ένα τομέα όπου εγώ ευθύ αμέσω, μόλι αναλάβω καθήκοντα, θα ε, στρέψω την προσοχή μου, διότι ήδη έχουμε αποφασίσει ότι η πρώτη μα αποστολή, η πρώτη μα επίσκεψη θα είναι στο Ελσίνκι, αν δεν κάνω λάθο, γιατί εκεί έχουμε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τα χημικά. Αυτό θα είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία έχουμε διακηρύξει. ε, αν με ρωτάτε αν είμαι ικανοποιημένο με, με τα όσα έχουμε αυτή τη στιγμή ως κείμενη νομοθεσία, θα σας πω όχι. I will use the technology of microphones. Um, the second part of the question was also on the definition of PBTs Ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Τι γίνεται με τα PBT, γιατί δεν καλύπτει η σύμβαση της Στοκχολμής όλα αυτά επίσης. Είναι δυνατόν να πιάσει κανείς πλακτόν με δίχτυα. Ε, τόσο ανεπαρκής είναι η κείμενη νομοθεσία. Οπότε αυτό που ζητούμε από εσά είναι να αναθεωρήσετε αυτή την κείμενη νομοθεσία που είναι ανεπαρκής. Ποτότσνικ. Σε τρεις ώρες θα το μάθουμε. Έχετε πρόβλημα με αυτά τα κριτήρια για τις ουσίες PBT. Τι να σας πω, θα ρωτήσω τον συνάδελφο Ταγιάννη τον νωρίτερο δυνατόν, τόσο να μπορέσουμε να πιέσουμε τα πράγματα για εξελίξεις. Και είμαι βέβαιος ότι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν με τον ε, σχετικό ορισμό τα προβλήματα αυτά κατά τη γνώμη μου είναι ότι γενικά όταν μιλούμε για οποιαδήποτε ουσία, δηλαδή για αυτέ που φέρνουν τι μεταλλάξει, για τα καρκινογόνα, όλα αυτά τα βιοσορευόμενα, όλα αυτά για τα PBT, όλε αυτέ τι ουσίε. Όποτε κανεί θέλει να το διερευνήσει θα πρέπει να μάθει ακριβώ περί τίνων πρόκειται. Πρόκειται για πάρα πολύ επικίνδυνε ουσίε. οπότε και εμεί θα πρέπει να ενεργούμε αναλόγω. Ε, Ευχαριστώ, Λέω πρόεδρο. Thank you. Um... Thank you. My question was also about implementation, which has been mentioned a couple of times, and your your answers were somewhat general, so I'm going to slightly change. my Απαντήσατε σε κάτι πρώτο πριν, ο... σε κάτι που με ενδιαφέρει, αλλά ήταν κάπως γενικό η απάντηση, οπότε εγώ επανέρχομαι. Τον Νοέμβριο του 2009 είχατε πει σε σχέση με τα απορρίμματα ότι θα πρέπει κάτι να γίνει για Κάτι θα πρέπει κάτι να γίνει για τη μη εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, κάτι θα πρέπει να γίνει για, όπου δεν υπάρχει ρύθμιση, κάτι θα πρέπει να γίνει για την παρόμοια απόρριψη των αποβλήτων. Είχατε ο ίδιος δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα το τι θα πρέπει τώρα να προσέξετε επομένως από πλευράς Κάποιο Ευρωπαίο πολίτη. Το ότι δεν έχει εφαρμοστεί το δίκαιο, αυτό σημαίνει ότι έχουμε αμφιβολίες και για την μελλοντική νομοθεσία κατά πόσο θα αποδώσει. Και ο πρόεδρος την κόβει. Uh, uh my, answer would be, uh, Ε, τώρα είναι αδύνατο να σας πω με λεπτομέρειες για το κάθε μέρος συγκεκριμένο ζήτημα. Ξέρω ότι έχουμε πολλά προβλήματα, έχουμε πολλές περιπτώσεις παραβιάσεων, έχουν 500-600 καταγγελίες ανά έτος και ότι έτσι έχει η κατάσταση εγώ. Θα κάνω ό,τι πρέπει από το χέρι μου. Ούτως ώστε να ισχύσουν όσα έχουμε εξαγγείλει και συμφωνήσει. Όμως από την άλλη μεριά θα πρέπει πάντοτε για το δεύτερο κομμάτι της πενταετίας μας να εκμεταλλευτούμε αυτό τα οποία μάθαμε το πρώτο μισό. Και αυτό το έμαθα από την προηγούμενη θητεία μου. Πάντα στην αρχή κανένας δεν είναι τόσο σίγουρος Άρα πρέπει να δούμε πώ θα πλουστεύσουμε την νομοθεσία, πώ θα την κάνουμε πιο ευφυή, πιο έξυπνη και με τίποτα δεν είπα να κατεβάσουμε τον πύχη των προσδοκιών. Όμω θα πρέπει να βάλουμε νομοθεσία η οποία να επιδέχεται εφαρμογή και η οποία να είναι απλή. Και έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για το περιβάλλον. Um, I, I Επερώτηση. Άλλο θέλω να μου πείτε και δεν μου το λέτε αυτό το οποίο περίπου κρυστεύει προηγουμένω, ότι δηλαδή θέλω να μα πείτε ότι έχετε δώσει υψηλή προτεραιότητα στο να μπορέσετε να κάνετε περισσότερα πράγματα όσον αφορά την εφαρμογή τη νομοθεσία σε σχέση με τα λίγα που έχουν γίνει στο παρελθόν. Άρα, φρένο στην καινούργια νομοθεσία μέχρι ότου εφαρμοστεί δεόντως η ισχύουσα. Higher on the agenda, it's a relative term, which means that it was not προτεραιότητα πάνω να πει ότι δεν υπήρχε πριν προτεραιότητα όταν ο συνάδελφος είχε την προηγούμενη θητεία. Εγώ σας υπόσχομαι ότι θα είναι ψηλή προτεραιότητα η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για μένα. Και θα το προσέξω αυτό το θέμα διότι πιστεύω ότι μόνο όταν εφαρμόζεται η νομοθεσία τότε έχουμε νομοθεσία που πραγματικά ωφέλει το περιβάλλον. Γιατί αν δεν εφαρμόσει κανεί νομοθεσία αυτή είναι άχρηστη. Όχι, όχι, δεν πρόκειται να έχουμε μορατόν, Δεν θα φρενάρω την θέσπιση νέας νομοθεσία, αλλά θα τα σκεφτώ καλά. Να έχουμε όσο γίνεται καλύτερη σχέση κόστο αποτελέσματο, να έχουμε όσο γίνεται λιγότερε αρνητικές συνέπειες, αλλά θα πρέπει, ε, όπως και να είναι, θα πρέπει να εφαρμόζει νομοθεσία και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η άποψή σας πρόκειται να προωθήσει την Ευρώπη στον ηγετικό ρόλο όσον αφορά την πολιτική των αηφορών πολιτικών. Ποιους μηχανισμούς έχετε εδώ κατά νου συγκεκριμένα. Θέλετε μια οικονομία οικολογικά υπεύθυνη με περισσότερους διακανονισμούς ή θα αφαιθείτε στην αγορά να διακανονιστεί μόνη της. Επιπλέον θα με ενδιαφέρε ποια είναι η απόψη σας για τη μεταφορά γνώσεων χωρίς ε, ευρυστεχνή στις αναπτυσσόμενες χώρες. That's for four in one. Uh, okay, I think uh, in essence we talk about an area which is internationally extremely connected. So, as I said in my introductory speak, σας τα είπα στην εισήγησή μου. Μιλάμε για παγκοσμιωμένο κόσμο, όλα είναι αλληλένδετα και επομένως και αυτό το οποίο λέτε οδηγεί σε ε, διεθνή συνεργασία που είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται. Επομένως, εμείς έχουμε δεσμευτεί σε σχέση με το πρόγραμμα του ΟΗΕ και για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο όργανο του ΟΗΕ και εκεί έχουμε εμπλακεί και δώσαμε και τις σχετικές δεσμεύσεις στο Ρίο, στην Κοπενχάγη για την αλλαγή του κλίματος και οπότε όλα αυτά δείχνουν το πόσο σοβαρά βλέπουμε το θέμα, πόσο βαθιά μας προβληματίζει Αλλά θα κινηθούμε σε αυτόν τον άξονα τη διεθνού, συνεργασία για θέματα του περιβάλλοντος και όταν αναφέρεστε στην νομοθεσία και σε μέσα πολιτικής που βασίζεται στην αγορά και τι προσεγγιστά έχουμε όλα αυτά εδώ τα έγγραφα που έχω είναι χειρόγραφα γι' αυτό σας τα λέω έτσι οπότε ολιστική προσέγγιση τι θα πει. Αν θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα είναι ότι χρειάζεται πολιτική πρωτοπορία, αποδοχή από το κοινό, ε, υποδομή, χρηματοδότηση, να λάβουμε υπόψη την αγορά, τιμολογική πολιτική, όλα αυτά, όλα, όλα μαζί χρειάζονται και αν συνδυαστούν όλα μαζί αποδίδουν. Σε μερικές περιπτώσεις αλλού δίνει λύση νομοθεσία και αλλού η αγορά. Εξαρτάται. Ολιστική προσέγγιση επομένω. Και έτσι μόνο μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα. Όλα τα άλλα είναι αβέβαιο αποτέλεσματο. Και για αυτόν τον τομέα τον κόβει ο πρόεδρο. Ja, ich habe jetzt verstanden, dass Sie der Regulierung keinen Vorrang einräumen. Ε, δηλαδή, θέλετε να δώσετε την προτεραιότητα στο διαγωνισμό και πώς προβλέπετε το μελλοντικό πρόγραμμα επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αηφόρο ανάπτυξη και για ε, θέσεις απασχόλησης που να έχουν μέλλον. Έχετε κάτι κατά νου για αυτού του είδους το πρόγραμμα. βέβαια και είναι προτεραιότητα η νομοθεσία και θα πρέπει να χρησιμοποιείται και όταν συζητήσαμε για τις εκπομπές του διοξιδίου από τα αυτοκίνητα, λέγαμε ότι χρειάζεται αυτή η νομοθεσία. Όμως από την άλλη μεριά είπε ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε την αυτοκινητοβιομηχανία. Αλλιώς βιαζόμαστε, τους τριμώχνουμε πολύ και μας χρειάζεται συνδυασμός του δημοσίου, του τομέα, τα προγράμματα ε, να χρησιμοποιηθούν τα κοινοτικά, να τους βοηθήσουμε κατά κάποια μεταβατική περίοδο. Όλα αυτά τα είπα και τα έκανα. Άρα χέρι-χέρι με τον ιδιωτικό τομέα. Να τους βοηθήσουμε ούτω ώστε να φτάσουν στο σημείο όπου δίνονται λύσεις που είναι και επικερδείς. Αυτό όμως δεν αλλοιώνει το πιστεύω μας ότι θα πρέπει να είμαστε αυστηροί στην νομοθεσία. Δηλαδή να έχουμε νομοθεσία αυστηρή αλλά προβλέψιμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάω σας ευχαριστώ πάρα πολύ πρόεδρε. Θα ήθελα αρχίζοντα να ευχηθώ σε όλους ευτυχές και κρύο νέο, νέο έτος. Φαίνεται ότι εγώ έμεινα από τους λίγους βουλευτέ. που δεν ε, αγριεύει όταν μιλάμε για την ε, ε αύξηση της του πολίτη που οφείλεται σε ανθρώπινες επεμβάσεις. Ας πάρουμε ε, λιγάκι το κοινό νου. Αν πάρουμε 100.000 χρόνια, που είναι λογικό για τις κλιματολογικές, 100.000 χρόνια, συγγνώμη, βλέπουμε ότι υπάρχει μια διακύμανση. Δεν πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή είναι υπερβολική, για να μην πω εγωιστική οι στάση αν λέμε ότι ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει το κλίμα. Ναι, μια που παλιότερα ήμουν υπεύθυνο για την έρευνα και την επιστήμη, ξέρω ότι ποτέ δεν συμφωνούν οι επιστήμονες για κάτι, αλλά σε έναν τομέα έχουμε ένα μέσο, είναι ακριβώς κλαματολογικές αλλαγές. Έχουμε ένα διεθνές βήμα για τις κλιματολογικές αλλαγές, όπου 600 περίπου επιστήμονες σε όλο τον κόσμο συμφωνούν. Ορισμένοι επιστήμονε βέβαια δεν συμφωνούν, το ξέρω, αλλά σε κανένα άλλο τομέα δεν έχουμε τόσου πολλού επιστήμονε που συμφωνούν. Η απάντησή μου θα είμαι κάπω προκλητική. Εάν, α πούμε, έχετε δίκιο, εσεί και εγώ δεν έχω δίκιο. Τι σημαίνει αυτό. Άλλε πολιτικέ που κάνουμε είναι σωστές. Είναι σωστό να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας όλους τους τομείς. Η απάντησή μου είναι ναι. Ακόμα λοιπόν και αν είναι λάθος αυτό, δεν συμφωνώ. Αλλά αν ήταν οι ίδιες πολιτικές θα πρέπει να ακολουθούν. Και το άλλο είναι, αν εγώ έχω δίκιο και εσείς έχετε ε, άδικο και ακολουθήσουμε τις ε, συμβουλές αυτών των κάποιων επιστημόνων, τι θα γίνει. Η απάντηση είναι σαφής. Καταστροφή. Ελπίζω ότι δεν χρειαστεί να φτάσουμε σε κάτι τέτοιο. Να μην έχουμε μια οικονομική κρίση, το ίδιο όπως είχαμε συγγνώμη στην οικονομική κρίση, που μάθαμε το μάθημά μας όταν έχει φτάσει η κρίση ήδη εδώ. Καλύτερα να αντιδράσουμε εκ των προτέρων. Όλα, τι έγινε με τις χιλιάδες εμπειρογνωμόνων που υπέγραψαν τη δήλωση του Ορεγκόν. Αλλά εντάξει. Εσείς καταστρέφετε την οικονομία επιβάλλοντας πράσινους φόρους, επιβάλλοντας τόσες διατάξεις. Και εδώ βασιζόμαστε σε τελείως φανταστικά μοντέλα στις υπολογιστές. Πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε μια τέτοια πολιτική η ε, μεθοδολογία και επιστήμη των ε, υπολογιστών μας έχει προχωρήσει. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι κανένας δεν θέλει οπωσδήποτε να εργαστεί ενάντια σε επιχειρήσεις. Εμείς θέλουμε η ε, επιχειρησιακή λογική να λάβει υπόψη κάτι που νομίζω πιστεύουν όλοι. Ότι θα πρέπει να περάσουμε σε μια νέα βιομηχανική επανάσταση του πρασινίσματος, της ενσωμάτωσης δηλαδή του κόστους του περιβάλλοντος. Απλό αυτό. Εάν στην αρχή αυτού του σκεπτικού μας ενσωματώσουμε το κόστος αυτών που χρησιμοποιούμε εμείς σαν καταναλωτές, πράγμα που θα πρέπει να γίνει, θα περάσουμε προς μια ανηφόρο κατεύθυνση. Αυτή είναι η απάντησή μου. Όσον αφορά στους διάφορους φόρους που αναφέρεται, οι κυβερνήσει θα μαζέψουν ό,τι φόρου θέλουν. Μην ανησυχείτε. Καλύτερα να τους ε, εισπράξουν από τους, για πράσινους λόγους ή για άλλους, αλλά τέλο πάντων. Πρόεδρος. Δεύτερος γύρος. Άνια Βάισκερ έχει την πρώτη ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Ποτός. και εγώ δεν θα αναφερθώ στην έλλειψη εφαρμογής αλλά στη διαφορετική εφαρμογή της ε, περιβαλλοντικής νομοθεσίας στα κράτη-μέλη. Γιατί θα πρέπει το περιβάλλον να προστατευτεί πέρα από τα σύνορα και να δημιουργήσει ενιαίες ε, προϋποθέσεις ανταγωνισμού στην Ευρώπη. Αλλά και οι δύο αυτοί οι στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν εάν οι οδηγίες εφαρμόζονται διαφορετικά στα διάφορα κράτη-μέλη. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα όπως η οδηγία για την ποιότητα του ατμόσφαιρας που όλα εξαρτάται από το ποια σημεία και πόσα σημεία ελέγχου θα υπάρχουν στα διάφορα ε, κράτη ή όταν υπάρχουν διαφορές ε, της τάξης του ε, παράγοντα χίλια μεταξύ των οριακών τιμών που ορίζονται. Είπατε κύριε ποτοτσιο ότι θα καταβάλλετε κάθε προσπάθεια για να εφαρμοστούν οι νομοθετικές διατάξεις. Τι θα κάνετε ούτως ώστε να μπορέσει να ελέγχει την εφαρμογή των οδηγιών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρχουν ενιαίοι όροι ανταγωνισμού. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ καλή ερώτησή σας. Γιατί είναι δύσκολη η απάντησή της. Και αυτό είναι κάτι που έμαθα εδώ. Ότι πραγματικά έχουμε ελλείψεις. Είναι καλό να έχουμε περισσότερες πληροφορίες ε, για τα, την εφαρμογή διαφορών οδηγιών. Ήδη έχουμε μία οδηγία του 2008 που προβλέπει κάτι τέτοιο και θα θέλω να την ενδυναμώσω. Και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για το Περιβάλλον στην Κοπενχάγη θα πρέπει να εργαστεί προς την κατεύθυνση αυτή και θα μελετήσω προσεκτικά τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Γιατί γνωρίζω ότι μόνο ε, όταν βασιζόμαστε καλά στις πληροφορίες μπορούμε να πάρουμε σωστές αποφάσεις. Όταν προετοιμάζουμε την νομοθεσία και εξετάζουμε όλες τις αναθεωρήσεις, αναθεωρήσεων που ξέρουμε όλοι, γνωρίζουμε όλοι, θα πρέπει να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη. Λοιπόν, ευφυής νομοθεσία, ίσο πεδίο παιδής και Σύνηση για να λάβουμε υπόψη μας τις περιφερειακές διαφορές όπου υπάρχουν πραγματικά καλά επιχείρηματα. Αυτό θα πρέπει να είναι τμήμα της λογικής μας και της ε, προσπάθειας του μέλλοντος. Ευχαριστώ. Ναι, τα προβλήματα του περιβάλλοντος ξεπερνάνε τα σύνορα και γι' αυτό υπάρχουν ε, ορισμένα βέβαια που πρέπει να λυθούν σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχουν άλλα που μπορούν να λυθούν σε επίπεδο εθνικό. Όπως παραδείγματο χάρη οι κανόνες που αφορούν τα εδάφη. Θα ήθελα να σα ρωτήσω εσείς προσωπικά ποια άποψη έχετε όσον αφορά τη συνέχιση της νομοθεσίας για την οδηγία προστασίας των εδάφων. Απάντηση. Εισαγωγικά, σας είπα ότι δεν θέλω η επικορικότητα να θεωρηθεί μια δικαιολογία για την αδράνεια. Από την άλλη μεριά θα τίσνω χέρι βοηθία σε όλα τα κρατημέλη για την εφαρμογή αυτή η οδηγία στην οποία αναφέρεστε η... προωθείται εδώ και πολλά χρόνια, το 2006 αν δεν κάνω λάθος. Θα πρέπει να δω πώς μπορεί να επιληθεί το θέμα στο Συμβούλιο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πέντε χώρες που είναι αντίθετες με την υιοθέτησή της. Δεν έχουμε δηλαδή την επαρκή πλειοψηφία για να εγκριθεί. Εγώ δεν θα αφαιρέσω την οδηγία αυτή για τα εδάφη από τη διαδικασία, γιατί είναι ένα θέμα ευρωπαϊκού συμφέροντος νομίζω. Πρόκειται για ένα τομέα, ένα τομέα που δεν καλύπτεται περπώς Ξέρω βέβαια ότι σε πολλά κράτη-μέλη εργάζονται πολύ καλά. Το ξέρω αυτό. Και ο στόχος της οδηγίας για τα τάφη είναι να μειωθεί αυτό. Ευχαριστώ. Ανδρέας Περέλιο Τρίγες. Πάρα πολύ χαίρομαι που συζητούμε σήμερα εδώ, αλλά έχω και μία ερώτηση. Είναι προτεραιότητά σα να συνεχθεί το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο για το περιβάλλον, κάτι το οποίο σήμερα, αυτό το χρόνο, πρόκειται να εκπνεύσει, να λήξει. Πρόκειται το συντομότερο δυνατόν να έρθει εδώ στο Κοινοβούλιο για να μα παρουσιάσετε το έβδομο πρόγραμμα για το περιβάλλον, το ευρωπαϊκό. Είναι κάτι το οποίο τώρα εκκρεμεί, μια όπου λύγει το έκτο. Επίση, για πέστε μα. υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με το τι θα κάνει η Κομισιόν. Άρα, προτίθεται η Κομισιόν να διασκεδάσει εκείνες τις εντυπώσεις, γιατί έγινε η Κοπενχάγη και με αυτά που γίνανε εκεί δεν είναι καιρός για αμφιβολίες. Εσείς δεσμεύεστε ενώπιόν μας ότι θα προχωρήσετε προς αυτή την κατεύθυνση. Thank you. Σας ευχαριστώ. Ε, 2002-2012 είναι η διάρκεια του έκτου περιβαλλοντικού προγράμματος δράσης. Προχωρούν τα πράγματα λοιπόν και θα έχουμε την αξιολόγηση του έκτου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον και προετοιμάζεται ήδη το λεγόμενο SOER που προετοιμάζει η αρμόδια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για το θέμα των, ε, της κατάστασης ε, του περιβάλλοντος στην Ευρώπη και τις προοπτικές για το μέλλον. Πρέπει να προετοιμαστούμε για τον Ιούλιο του 2012. Αλλά εσύ μας ρωτήσατε τι έχω κατά νου για το 7ο πρόγραμμα. Αν ακολουθήσω τη γραμμή που έχει αναφερθεί εκεί στην προετοιμασία, ξέρετε ποια θα είναι η απάντησή μου τυπικά εγώ δεν μπορώ να δεσμευτώ γιατί υπάρχουν διάφοροι διακανονισμοί που θα πρέπει να καθοριστούν, να διευρυθούν κλπ. Αλλά κοιτώντα αυτό το θέμα τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το 2012 και μετά τη στρατηγική της ε, φόρου ανάπτυξη, που νομίζω αφορά το, την Ευρώπη 2020, Πιστεύω ότι το έβδομο πρόγραμμα δράσης θα πρέπει να είναι ιδανική δυνατότητα να εξεταστούν διάφορα από τα θέματα εις βάθος. Και ε, το να περάσει αυτό σε διαδικασία συναπόφασης για μένα είναι πλεονέκτημα, γιατί έτσι θα μπορέσουμε αναλυτικά να εξετάσουμε τα θέματα που θα μας απασχολούν στο μέλλον. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν είναι επίσημη δέσμευση, αλλά νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να σας ικανοποιήσει. Ωραία. Και εμεί ελπίζουμε αυτή σας ειδική δέσμευση να υλοποιηθεί. Για την ατμόσφαιρα τώρα. Σε κάποια κράτη έχουμε τόσο χαλαρή νομοθεσία που σε κάποιε πόλει δεν γίνεται τίποτα για να βελτιωθεί η ποιότητα. Και οι μετρήσει είναι άλλα αντάλλων, ανάλογα με τον τόπο όπου γίνονται. Άρα θα πρέπει να πιέσετε τα κράτη-μέλη να κάνουν περισσότερα. Εσείς θα θεσπίσετε τα αντίστοιχα νομοθετήματα ούτως ώστε να τραβήξουμε το λουρί σε αυτούς που έχουν χαλαρή νομοθεσία. Στα όρια. Στα όρια των κανόνων. Είναι μάλλον μια δεύτερη ερώτηση. Δεν θα την εγκρίνω. Θα περάσουμε στον επόμενο. Ε... Ο κύριος Κράμερ έχει το λόγο. Κύριε υποψήφια επίτροπε, ας με απασχολεί το θέμα της δημοκρατίας και της πυκνότητας των διακανονισμών, γιατί έχουμε πάρα πολλή νομοθεσία που δεν πληρεί το ρόλο της, αλλά δημιουργεί περισσότερη γραφειοκρατία. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι στις πρωτοβουλίες που θα υποβάλλετε τα επόμενα χρόνια θα έχετε κατά νου το θέμα της αποτελεσματικότητας των δαπανών ε, περισσότερο από ότι ο προκατοχός σας και θεωρείτε να υπάρχουν κάποιοι τομεί τη περιβαλλοντική πολιτική όπου μπορούμε να σταματήσουμε με τον διαγωνισμό όχι για να έχουμε λιγότερη προστασία του περιβάλλοντος αλλά για να μπορέσουμε να προφτάσουμε να εφαρμόσουμε αυτά που έχουν ήδη υιοθετηθεί. Στις αξιολογίες επιπτώσεων θα πρέπει να εξετάζουμε πάντα την περιβαλλοντική διάσταση. Θα πρέπει να ε, τα έχουμε όλα αυτά κατά νου. Πολύπλοκη νομοθεσία, ακριβή νομοθεσία, που ξέρουμε εκ μιας αρχής ότι δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί, δεν είναι προ όφελο ουδενός. Οπωσδήποτε δεν είναι προ όφελο του περιβάλλοντος. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να εξτάσουμε όλες τις δυνατότητες. Ο ρόλο μα είναι να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Πρώτο και κύριο. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να το πετύχουμε αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε διάφορου τομεί. Απλούστευση όμω είναι ένα από τα θέματα όπου είμαι λιγότερο ικανοποιημένος αυτή τη στιγμή. Προσπάθησα να κάνω ό,τι μπορούσα. Έκανα κάθε μέρα ό,τι μπορούσα για να πιέσω προς την κατεύθυνση αυτή. Το μόνο που μπορώ να πω είναι στο τέλος της ε, θητείας οι όροι είναι τέτοιοι που ο διάδοχός μου έχει τις ειδικές προϋποθέσεις για απλούστευση της έρευνας, γιατί είναι τώρα πολύ γνωστό αυτό το θέμα και γνωρίζετε απόλυτα τι πρέπει να ε, αλλάξει και τι όχι. Σας το εξηγώ αυτό για να καταλάβετε δηλαδή την κύρια μου σκέψη στον τομέα αυτό. Νομίζω ότι εφής ε, νομοθεσία, απλούστευση κλπ να μην έχουμε πολύ γραφειοκρατία είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ότι εδώ εγώ είμαι υπεύθυνο για το περιβάλλον. Είμαστε εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουν τα πράγματα να προχωρήσουν αηφόρα στο μέλλον. Ένα παράδειγμα για κάτι που προωθείται αυτή τη στιγμή είναι η πολιτική για τις βιομηχανικές εκπομπές, διακόπτει ο Πρόεδρος. Herr Kommissar, kann ich Sie darauf festnageln, dass kein Gesetzesvorschlag hier... Κοιτάξτε, θα ήθελα να σας πω τι θα γίνει όσον αφορά τις, την αξιολόγηση των επιπτώσεων, κατά τη γνώμη σας. Yes, I think that's the correct way. Ναι, νομίζω πως αυτό είναι ο σωστός τρόπος. Ότι κάθε δηλαδή νομοθεσία θα πρέπει να περνά από μια εξονυχιστική αξιολόγηση αντικτύπου και το περιβάλλον θα πρέπει να είναι πάντοτε παρόν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υποψήφιο Επίτροπε, το ερώτημά μου αφορά την βιοπικιλότητα που την αναφέρατε και εσείς ως προτεραιότητα και που πιστεύω ότι είναι προτεραιότητα και του δικού μας σώματος. Η προστασία της βιοποικιλότητας χρονολογείται από το 2000 με τη σχετική νομοθεσία. Πάνω από 120 διαδικασίες παραβίαση έχουν ξεκινήσει κατά των διαφόρων κρατών μελών γιατί πολλά από αυτά έχουν ανεπαρκώς εφαρμόσει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τα κράτη-μέλη αυτά βεβαίως θα πρέπει να τιμωρηθούν. Αλλά, αλλά επειδή τα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα οι περιφέρειες αγωνίζονται με κάποια στοιχεία αυτής της νομοθεσίας, για παράδειγμα των αόριστους ε, ορισμούς, ε, ε, η νομοθεσία, όπως είπαμε, ε, ε, χρονολογείται από το 1979 και δεν λαμβάνει υπόψη τι κλιματικέ αλλαγέ, ε, τουλάχιστον όπως τις γνωρίζουμε σήμερα. Προτίθεστε να ενημερώσετε την νομοθεσία περί βιοποικιλότητας θα, είτε δίνοντα προτάσει είτε περισσότερε κατευθύνσει προ τα κάτι μέλη, αποσαφηνίζοντα ας πούμε αυτού του ορισμού, είτε διαδίδοντα τι καλύτερε πρακτικέ. Αυτά. Η απάντηση αφορά περισσότερο το δεύτερο κομμάτι της ερώτησής σας. Ε, σκοπεύω να ακολουθήσω αυτή την κατεύθυνση, ε, να είμαι πιο συγκεκριμένος. Νομίζω πως ε, η βιοπικιλότητα είναι πολύ σημαντικό θέμα. Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά από πράγματα δηλαδή πρέπει κανείς να λάβει υπόψη. Το ένα βεβαίως αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας όταν Κάποιες φορές η νομοθεσία είναι πολύ ξεκάθαρη, το Natura είναι πολύ ξεκάθαρο, φορά τα, τους οικοτόπους. Η Σλοβενία έχει 35,5% του εδάφους τους της στο Natura, για να ξέρετε πού βρισκόμαστε. Είναι πολύ καλό διατηρημένη χώρα. Είναι σημαντικό όταν εξετάζουμε τα θέματα της εφαρμογής λοιπόν να εφαρμόζεται με τον τρόπο με τον οποίο είχε προβλεφθεί από την αρχή της σύνταξης νομοθεσίας. Ό,τι γίνεται στις περιοχές Natura γίνεται με την πρόθεση να προστατευτεί η φύση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι καμιά από τις δραστηριότητες σε αυτή την περιοχή δεν επιτρέπεται. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν καλά παραδείγματα, όπως είπατε και εσείς, που θα πρέπει να τα δούμε και να τα ακολουθήσουμε και σίγουρα εγώ σκοπεύω να ακολουθήσω αυτή την κατεύθυνση, ότι δηλαδή τις γνώσεις που έχουμε από τα καλά παραδείγματα να τις ε, εκμεταλλευτούμε και έπειτα θα, ε, μετά από επισκέψεις στην Ολλανδία και τη Γερμανία για παράδειγμα ε, είδα ότι τα περισσότερα παραδείγματα Ε, κακής εφαρμογής και κακών ε, ε, συναισθημάτων προέκυψαν λόγω ακριβώς της εφαρμογής αυτών των προγραμμάτων και είδα πού έγκυται το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ που εγινε το προβλημα τόσο δραστήρια προσέγγιση. Τώρα, αν δεν τα καταφέρουμε το 2010, αν βάλουμε στόχο το 2015, ποια θα ήταν τα βασικά θέματα που θα πρέπει να αλλάξουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτευχθεί ο επόμενος μας στόχος το... για τη βιοπικιλότητα Αυτή τη στιγμή, για την πρώτη ερώτηση απαντώ ακόμα, δεν, ε, δεν έχω πρόθεση να αλλάξω την ίδια την νομοθεσία. Η, αλάτηση, η ερώτηση που μας, ε, μου κάνετε τώρα, ειδού η απάντηση. Καταρχήν, ε, εφαρμογή της νομοθεσίας όπου έχουν καθοριστεί οι περιοχές θα πρέπει να επιταχυνθεί η εφαρμογή ή μάλλον ο καθορισμός των περιοχών. Δηλαδή η πρώτη απάντηση είναι η εφαρμογή, μετά έχουμε κενά και για τα εδάφη και για τα είδη. Τρίτον είναι να βελτιωθούν οι γνώσεις μας. Έχουμε έλλειψη γνώσης, έχουμε έλλειψη όσον αφορά την καταμέτρηση, έχουμε βεβαιότητες ως προς την αξία της βιοποικιλότητας, το κόστος, δηλαδή και ο κίνδυνος της βιοαπόλειας δεν είναι, δεν είναι σαφές και έπειτα και πάλι εδώ θα πρέπει να έχουμε περισσότερο ολιστική προσέγγιση να εφαρμόσουμε αυτή τη λογική για την κοινή γεωργική πολιτική και για την κοινή αλλιευτική πολιτική. Ähm, Κύριε είμαστε όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σαν Επιτροπή οι ηγέτες στον τομέα του περιβάλλοντος και αυτό είναι για πολλούς Ευρωπαίους και Ευρωπαίες ένα μεγάλο πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ακριβώς στον τομέα αυτό είμαστε εκείνοι που προηγούμε σε όλη την υφήλια. Από την άλλη μεριά έχουμε συνεχώ δυσκολίε να κοινοποιήσουμε αυτά τα πλεονεκτήματα και έχω εδώ κατά νου την κατάσταση που είχαμε με την απαγόρευση των παλιού τύπου λαμπτήρων. Πώς σκέφτεστε, πώς θα μπορούσε να παρουσιάσετε στους πολίτες της Ένωσης ε, τις, ε, τα επιτεύγματα που θεωρητικά τα θέλουν οι πολίτες αλλά δεν τα θέλουν πρακτικά. Ποια θα είναι η πολιτική σας επικοινωνία που θα ακολουθήσετε. Again, not an easy Και πάλι δύσκολη ερώτηση. Νομίζω πως ε, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι να καταλάβουμε όταν συζητάμε τα θέματα αυτά ότι ό,τι και αν κάνουμε πρέπει να το κάνουμε έχοντας υπόψη πως δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο το αύριο, αλλά είναι κάτι μακροπρόθεσμο. Η μακρο, δηλαδή, το, το μακρόπνο όραμα δεν λαμβάνεται αρκετά συχνά υπόψη νομίζω. Και αυτό είναι επίσης σημαντικό όταν λαμβάνονται τέτοια μέτρα. Γιατί και όταν ασχολούμαστε με θέματα τα οποία δεν είναι αναστρέψιμα. Γιατί η ζημιά τότε έχει ήδη γίνει και δεν μπορεί να διορθωθεί. Το να επικοινωνούμε βέβαια με τον κόσμο και να ενημερώνουμε αρκετά, αλλά να έχουμε και την άποψή του είναι πάντα δύσκολο. Αλλά Καλύτερο τρόπος για να επικοινωνούμε με τον κόσμο είναι οι καλές πολιτικές και οι σωστέ αποφάσει. Ε, θα πρέπει δηλαδή να προσπαθούμε να, ειλικρινά να εξηγούμε και να μην καταχρώμεθα. Τις νομοθεσίες. Πρέπει να είμαστε δηλαδή έντιμοι, ειλικρινείς και να εξηγούμε για το ότι δεν υπάρχουν άλλο είδους συμφέροντα, είτε περιφερειακά είτε επιχειρηματικά, αλλά ότι πραγματικά πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε. Αυτή ε, ε, βέβαια η καλύτερη πολιτική προϋποθέτει και την καλύτερη μέθοδο εφαρμογή. Απ' την άλλη μεριά όμως θα πρέπει να ασχοληθούμε με τους διάφορους ενδιαφερόμενους. Αν σκεφτώ παραδείγματος το θέμα του ανταγωνισμού, όταν έχουμε μέτρα περιβάλλοντος που από πλευρά επιχειρησίων ε, υπάρχει εντύπωση ότι περιορίζουν την ανταγωνιστική του δυνατότητα. Απ' την άλλη μεριά όμως είναι προς όφελος των καταναλωτών. Πώς μπορείτε να συνενώσετε εσείς τα δύο αυτά. Όχι μόνο ο κόσμος, αλλά και ο επιχειρηματικός κόσμος θα πρέπει να καταλαβαίνει. Νομίζω πως ε, αυτή η συνεννόηση ωστόσο γίνεται και πιο προφανής ε, καθημερινά. Πάντως δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να θεωρήσουμε αυτονόητο. Ωστόσο, εάν όλοι πραγματικά είμαστε συνεπείς αν είμαστε συνεπείς στην παροχή επιστημονικών στοιχείων, αν είμαστε συνεπείς στο να γνωστοποιούμε και να τεκμηριώνουμε τα όσα αποφασίζουμε και θέμα να αποφασίζουμε, τότε το κοινό σίγουρα θα τα καταλάβει καλύτερα. Στα περιβαλλοντικά ζητήματα νομίζω πως είμαστε πολύ ανοιχτοί και ειλικρινείς και γι' αυτό και αν δείτε το ευρωβαρόμετρο για το πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος όλα αυτά τα θέματα, η κατανόηση είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Νομίζω πως είμαι ανάμεσα στα, στους λίγους τυχερούς που έχουν ασχοληθεί με τομείς που είναι πολύ εύληπτοι για τον, άνθρω... για τον κόσμο, δηλαδή περιβάλλον και ε, έρευνα και ανάπτυξη. Μερικά έξτρα δευτερόλεπτα λοιπόν, γι' αυτό θα κερδίσετε. κύριος Άντερ, Γιάννος Άντερ. Η καταπολέμηση της διασυνοριακής ρήπανσης είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία στο οποίο θα πρέπει να ληφθούν αυστηρά μέτρα στο άμεσο μέλλον. Ελπίζω πως θα συμφωνεί ο υποψήφιος επίτροπος μαζί μου. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πριν 10 χρόνια μία επιχείρηση αυστραλοκαναδική που δρούσε στην Ρουμανία σε ένα χρυσορυχείο μόλυνε, ρήπανε ε, με κιάνιο το ποτάμι που περνούσε δίπλα. Οι ζημιές ήταν τεράστιες ε, τόσο για τον κόσμο που κατοικούσε δίπλα όσο και για την οικονομία της χώρας. Αυτή τη στιγμή έχουν περάσει 10 χρόνια και κατασκευάζονται νέα ε, χρυσορυχεία που χρησιμοποιούν εκ νέου αυτή τη τεχνολογία του κιανίου. Μα αυτή η τεχνολογία θα έπρεπε να έχει απαγορευτεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Διερωτώ με λοιπόν και έχει γίνει αυτό και στην Ουγγαρία και στην Τσεχία εξάλλου ο υποψήφιος επίτροπος συμφωνεί και υποστηρίζει αυτή μου την φιλοδοξία. Nature and the consequences of the pollution Αναφέρατε ένα μόνο από τα προβλήματα. Όταν οι επιπτώσει τη ρήπανση είναι διασυνοριακέ, έχουμε νομίζω μεγαλύτερο πλεονέκτημα, γιατί μπορούμε να δούμε το θέμα αυτό και από την άποψη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να έχουμε μια κοινή άποψη και κοινή προσέγγιση. Φυσικά, είναι σαφές ότι από την άποψη της, την πλευρά της Κομισιόν οφείλουμε να σεβαστούμε τις τα νόμιμά μας όρια και δυνατότητες. Για παράδειγμα, όταν, κάνουμε, όταν έχουμε την οδηγία για την αντίκτυπο στο περιβάλλον, έχουμε και την οδηγία, την SEA, και νομίζω πως Οποτεδήποτε προσεγγίζουμε οποιαδήποτε πρόγραμμα ή σχέδιο, θα πρέπει να επιμένουμε ώστε τα συγκεκριμένα τμήματα της οδηγίας να εφαρμόζονται. Κατ' ουσίαν λοιπόν συμφωνώ μαζί σας, αλλά θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι οφείλουμε να ακολουθήσουμε τις ε, νόμιμα συμπεφωνημένες οδηγίες. Ορισμένα πράγματα εξαρτώνται από τα ίδια τα κρατημέλη, ενώ ορισμένα άλλα πρέπει να εφαρμοστούν στο επίπεδο τους. Όταν όμως υπάρχουν διασυνοριακές επιπτώσεις, είναι σκόπιμο να εξετάζονται οι υποθέσεις αυτές και από μια άλλη προοπτική. Ε, εγώ διαμαρτύρομαι εναντίον της δικής σας θέσης. Υπάρχουν κανόνες φυσικά. Αυτοί οι κανόνες ωστόσο εδώ και δέκα χρόνια δεν μας βοηθούν να λύσουμε το πρόβλημα. Άρα το θέμα δεν, βρει, δεν είναι η, η ισχύουσα νομοθεσία, είναι οι νέοι κανόνες, νέα νομοθεσία, πλήρης απαγόρευση χρήσης αυτής της τεχνολογίας, γιατί ο κίνδυνος ανανεώνεται διαρκώς αυτή η εξορυκτική τεχνολογία με τη χρήση κενίου θα πρέπει να απαγορεύεται παντελώς. Αυτή μόνο είναι η λύση. Γιατί διαφορετικά για τους υδροφόρους ορίζοντάς μας, για τους οριζόνες μας και για τον κόσμο που ζει εκεί γύρω είναι τρομερός ο κίνδυνος. Δεν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας τότε. Εάν δεν υπάρχει κατάλληλη οδηγία και αν υπάρχει σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα, το οποίο είναι προφανέ, φυσικά και θα πρέπει να το εξετάσουμε. Εάν απαιτείται απαγόρευση, θα απαγορευτεί. Αυτή τη στιγμή, θα, θα έλεγα δηλαδή ότι αυτή είναι η κεντρική μου θέση, αλλά μάλλον κατάλαβα λάθος την ερώτησή σας. Νόμιζα πως η, ερώτησή σα ήταν γενικότερη. Δεν κατάλαβα ακριβώ τι εννοούσατε. Πάντως η βασική μου ερώτηση είναι ότι Εφόσον δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία και υπάρχει σοβαρός περιβαλλοντικός κίνδυνος, φυσικά και θα πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Εξάλλου, είστε παρόν εδώ ε, και η φωνή σας εισακούγεται. Ε, από μένα εξαρτάται να προσπαθήσω να δω από τη δική μου πλευρά, να συγκεντρώσω στοιχεία, να καταλάβω τι συμβαίνει και να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ερχόμαστε στον τρίτο γύρο ερωτήσεων και πρώτος είναι ο Γκαστόν Φρανκό από το ΕΛΚΑ. Please. Merci, Σας ευχαριστώ κύριε υποψήφιε επίτροπε. Μιλήσαμε για το νερό, για τον αέρα. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για τα δάση. Είστε έτοιμος κύριε Επίτροπε να στηρίξετε τη δημιουργία μιας ε, πραγματικής ε, ολοκληρωμένης δασικής πολιτικής για την Ευρώπη. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να προωθήσετε την βιώσιμη διαχείριση των δασών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για να ενθαρρύνετε μια αποτελεσματική και καλύτερη κινητοποίηση των φυσικών πόρων, ιδιαίτερα του, της ξυλίας και της βιομάζας σκοπεύετε να φτιάξετε ένα κριτήριο βιωσιμότητας για τη βιομάζα. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να το καλύψω όσο γίνεται καλύτερα. Για μένα, τα δάση αποτελούν τμήμα μιας πολύ κρίσιμης ερώτησης. 30% της απασχόλησης και 40% της ε, γης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των εδαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνδέονται πολύ με τις κλιματικές αλλαγές. Παίζουν καθοριστικό ρόλο τα δάση. Νομίζω πως μέχρι σε αυτό το σημείο όλοι συμφωνούμε. Υπάρχει ένα θέμα ότι διεθνώς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατευτούμε κατά της αποψήλωσης των δασών. που σκοπεύουμε να κάνουμε εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, γνωρίζετε ότι υπάρχει το λευκό βιβλίο για την προσαρμογή στι κλιματικέ αλλαγέ από τον Απρίλιο του 2009, είναι υποσυζήτηση. Το πράσινο βιβλίο, το οποίο προετοιμάζεται για την προστασία των δασών ε, θα το λάβετε σύντομα. Είναι δύο πράγματα που είναι τα πιο σημαντικά για μια επικοδομητική και ευρεία συζήτηση μέσω της οποίας θα πρέπει να κατανοήσουμε σαφώς το πώς θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ή να ενημερώσουμε την, ε, να ανανεώσουμε μάλλον την στρατηγική της Ένωσης Περιδασών, καθώς και να διευκρινίσουμε και να απαντήσουμε στα ερωτήματα για το κατά πόσο η οδηγία πλαίσιο για τα δάση είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε ή όχι. Επίσης, ε, ένα συνεπές σύστημα για την ενημέρωση για τα δάση, για πληροφόρηση για τα δάση είναι σημαντικό. Je vous remercie, monsieur le... Σας ευχαριστώ κύριε υποψήφιο επίτροπε. Πιστεύω πως η απάντησή σας ε, δείχνει πως ε, έχετε όντως συνειδητοποιήσει τη σημασία του θέματος. Επίσης, ε, θα προσέξω ιδιαίτερα την ε, υιοθέτηση μέτρων που στόχο θα έχουν την επαλήθευση το, της, του σεβασμού των αποφάσεων που θα λάβουμε και κυρίως η καταπολέμηση της αποψήλωσης των δασών. Uh, Έχω ένα λεπτό για να επαναλάβω ε, αρκετές φορές ναι, ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Ιδιαίτερα από διεθνή άποψη θα πρέπει να παίξουμε το ρόλο μας εντατικά. Προέκυψαν και διάφορες συνέπειες μετά την Κοπενχάγη όπου σαφώς ε, συμφωνήθηκαν κάποια μέτρα για την διεθνή προσέγγιση. Ένα από τα ερωτήματα που συνδέονται με αυτά είναι και η χρηματοδότηση. Από την άλλη πλευρά αυτό που θέλουμε και πρέπει να κάνουμε, και αυτή είναι νομοθεσία που ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή, και παράνομη υλοτόμηση, μέσω μιας νέας προσέγγισης εδώ προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι γίνεται. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα με το ΦΛΕΚΤ. Έχουμε μια συμφωνία με την ΚΑΝΑ, όπως γνωρίζετε είναι η πρώτη διμερή συμφωνία και αυτό είναι καλό. Και αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο σκοπεύουμε να προχωρήσουμε. Όμως υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί σε όλα αυτά. Και νομίζω πως ναι, θα πρέπει εδώ να είμαστε πολύ, πολύ επιμελείς. Ευχαριστώ πολύ ο Βικτόριο Πρόντι. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. να χαιρετήσω τον Επίτροπο Ποτόσνικ με τον οποίο συνεργαστήκαμε πολύ καλά για την έρευνα κατά τη διάρκεια της περασμένης ε, θητείας της Κομισιόν. Ε, πολύ, πολύ ευπρόσδεκτες είναι τα όσα είπατε για το έδαφος και για την ανάγκη να ξαναδούμε την οδηγία γιατί προφανώς ε, καθίσατε όλο ένα και σαφέστερο ότι το έδαφος είναι εξαιρετικά σημαντικό ως απόθεμα, όπως μάλλον ε, αποθηκευτικός χώρος για τον άνθρωπο και ε, νομίζω λοιπόν ε, ότι το πιο σημαντικό τώρα είναι οι προσαρμογές στις κλιματικές αλλαγές που θα πρέπει να περάσουν μέσω της ολοκληρωμένης διατήρησης των εδαφών και άρα ιδιαίτερη προσοχή που θα πρέπει να δοθεί στα εδάφη και ήθελα να ακούσω ποια είναι η δική σας αντίδραση σε σχέση με αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα να σας πω ότι και εγώ αυτά πιστεύω για αυτά που κάναμε στο παρελθόν ε, και ακριβώ, ε, γι' αυτό και το πολύ επικοδομητική αυτή πενταετία. Τώρα σαν πρώτο έδαφος ε, σας είπα τι θα κάνω και συμφωνώ 100% με την ανάλυση για το πόσο σημαντικά είναι αυτά που είπατε από όλες τις πλευρές τώρα όσον αφορά για, την, τον συντονισμό, για την αλλαγή του κλίματος η συνάδελφος Χέντεγκρατ η Κόνη αντιγραφή θα το αναλάβει. Όμως θα, πρέπει να, τα πούμε στις λεπτομέρειες και πρέπει να σου πω ότι οτιδήποτε αφορά χαρτοφυλάκιο άλλου συναδέλφου είναι κάτι το οποίο αφορά το σύνολο της Επιτροπής. Αυτά έχουν οριστεί. Εγώ στο χαρτοφυλάκιο μου έχω το θέμα του περιβάλλοντο. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια είναι θέμα περιβάλλοντο. Μόνο εγώ θα το φροντίσω. Επομένω, εγώ σα εξηγώ από δική μου οπτική γωνία τι ισχύει. Εγώ επομένω θα καλύψω ό,τι μπορώ να καλύψω και θα φροντίσω το ώστε να να, να φροντίσουμε η βιοπικιλότητα, το έδαφος, το, το, το, το, το νερό, όλα αυτά, ό,τι μπορεί να κάνει η Γενική Διεύθυνση για το περιβάλλον. Αυτή την ευθύνη αναλαμβάνω και γι' αυτό δεσμεύτηκα όταν προτάθηκε αυτό το αξίωμα. Ε, με αυτό ήθελα να επανέλθω. Γιατί έχω την αίσθηση ότι υπήρχε ένας ε, κατακαιρματισμός εντολών και άρα είναι πολύ δύσκολο, ακόμα και για μας εδώ, Γιατί ο επίτροπος πούμε, που προτείνεται για την διεθνή εκπροσώπηση, την, ανθρώπινη, την ανθρωπιστική βοήθεια και την αντιμετώπιση των κρίσεων είπε ότι κατά κάποιο τρόπο η πρόληψη των ε, φυσικών καταστροφών είναι στη δική του αρμοδιότητα. Εγώ ανησυχώ λοιπόν πάρα πολύ γι' αυτό. Και εν πάση περιπτώσει ήθελα το σχόλιο σας. Uh, Μπορώ να σας πω τα εξής. Ότι στην Επιτροπή θα πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό το οποίο προσπαθούμε να καταφέρουμε από κοινού είναι ένα αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα αντίστοιχο με τις προσδοκίες σε σχέση με το τι πρέπει να κάνουμε. Και αυτό αφορά και τις δικές σας προσδοκίες. Ε, έχουμε πάρα πολλά νομοθετήματα που στο παρελθόν ήταν πρωτοβουλία περισσότερων του ενός επιτρόπων. Πολλές τέτοιες περιπτώσεις είχαμε και θα έχουμε και στο μέλλον. Άρα, πρόκειται να υπάρξει ευρεία συνεργασία για το οποίο μου αρέσει. Άλλωστε αυτό Έγινε και στο παρελθόν όπως είπατε και εσείς και είχαμε ένα σωρό περιπτώσει συνεργασιών και με την κυρία Χέντεγκαρντ επίση θα είπαμε για το πώ θα οργανώσουμε την συνεργασία μα για το μέλλον. Συνεργασία. Και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει κανεί ότι εγώ έχω προτείνει να έχουμε κοινέ συναντήσει των γραφείων των δύο επιτρόπων. Και ακριβώ γιατί είναι τόσο σημαντικό το να υπάρχει συνεργασία. Ευχαριστούμε λέει ο κύριος Γκέρμπραντι, για τις τόσο ξεκάθαρες ευθείες απαντήσεις. Ε, και εγώ θέλω να μιλήσω για την βιοποικιλότητα. Με ικανοποιείτε ότι για σας είναι το υπερθμόν δύο σπουδαίο ζήτημα που αντιμετωπίσετε και θα αναλάβετε να εικονίσετε μια καινούργια στατική για την βιοποικιλότητα. Στο παρελθόν, μάλλον σε αυτό τον ε, τομέα, αν θέλουμε να είμαστε πρέπει να πούμε ότι έχουμε αποτύχει, ότι αποτύχαμε. Οπότε, νομίζω ότι ο μόνος τρόπος να μπορέσουμε να πετύχουμε είναι εάν συσσωματώσουμε το κόστος της χρήσης των φυσικών πόρων στην ε, οικονομία μας. Οπότε, σας ρωτώ, εσείς θα το προσέξετε αυτό όσον αφορά τη νέα στρατηγική που θα χαράξετε. Δεύτερη ερώτηση. Τι θα κάνετε όσον αφορά το να πείσετε τους αδέλφους, ας πούμε, για την γεωργία, για την αλία, σε σχέση με το πόσο σημαντική είναι η Πάρα πολύ δύσκολο αυτό, λέει ο Επίτροπος. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι σε σχέση με το στόχο του 2010, στο παρελθόν όντως δεν τα πήγαμε καλά και αυτό είναι αρκετά κατηγορηματική διαπίστωση για να κάνουμε μια νέα προσέγγιση, γιατί ακριβώ ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε τη βιοποικιλότητα. Πρόσφατα υπήρξε αυτή η ανακοίνωσή μα που αφορά το νέο πρόγραμμα δράση για την ε, βιοποικιλότητα. Με το έτος του 2010, τέλος του 2010 θα το έχουμε ε, ξεκαθαρίσει, το έχουμε εκπονήσει. Ε, με το θέμα με απασχολεί. έχουμε κάποια κένα στη γνώση μας, στην πληροφόρηση, εκεί θα πρέπει να δουλέψουμε εντατικά. Και από πλευράς οικονομίας, και αυτό θα ληφθεί υπόψη, Πάντως, κατά τη γνώμη μου, η ουσία είναι ότι άπαξε κινούμεθα σε οικονομία αγοράς, το κόστος της κάθε πολιτικής θα πρέπει να ενσωματώνεται, να μετακυλίεται στο τελικό προϊόν. Αν αυτό υλοποιείται, τα πράγματα γίνονται πιο απλά. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, τότε κανένας προχωράει στο ράβε ξύλων. Μία λάθος απόφαση να και μετά έχουμε άλλα δέκα διορθωτικά μέτρα. Επομένω, αυτέ εξ αρχή θα πρέπει να ξεκινάμε το δεξί. Τώρα, όσον αφορά τον τρόπο τη συνεργασία, κοινή ερωτική πολιτική, κοινή αλληλευτική πολιτική, τα διευθυντικά ταμεία, τα δάση, όλα αυτά. Όλα αυτά είναι σημαντικοί παράγοντες για τη βιοποικιλότητα. Και όταν λέμε για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές, έτσι θα προσεγγίσω τους αρμόδιους συναδέλφους και έτσι θα προχωρήσουμε προς την συνεργασία επέκρινε ο Ολλανδός Πρωθυπουργός την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε σχέση με το περιβάλλον. Και δεν είπε ότι αντιτίθενται στα δικά του σχέδια αυτά που λέει η Ευρώπη, αλλά είπε ότι ο κόσμος δεν στηρίζει αυτή την ευρωπαϊκή πολιτική. Εσείς τι θα κάνετε, ούτως ώστε να ξανακερδίσετε τους Ευρωπαίους και τελικά να στηρίξουν την ε, περιβαλλοντική πολιτική. Ποτότσινικ. Να μην ξεχνούμε όσο αυτή την νομοθεσία το ότι εκπονείται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίνεται και επιψηφίζεται από Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Δεν είναι λοιπόν κάτι που κατεβαίνει έτσι ξαφνικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι κάτι που του έχει όλου σύμφωνου. Και αυτό προβλέπει και η συνθήκη. Και θα πρέπει έτσι να εφαρμοστεί σε αυτή η νομοθεσία. Βεβαίω υπάρχουν και συγκεκριμένε περιπτώσει, θα πρέπει κανεί να τι βλέπει διαφοροποιημένα. Και εμένα με απασχολεί το τι θα γίνει στι ε, κάτω χώρε Να δούμε ποιο είναι το πραγματικά το πρόβλημα εκεί. Και όσον αυτό το μήνυμα πρέπει να στείλει κανεί στον κόσμο, πιστεύω ότι είναι δύσκολο κανεί να ανταγωνιστεί, εδώ από τις Βρυξέλλες, να ανταγωνιστεί το εθνικό πολιτικό κλίμα. Είναι επομένω ευθύνη των αρμοδίων των πολιτικών στα κράτη-μέλη. Να λαμβάνουν και αυτοί το, το τη της ευθύνη σου για όλα αυτά τα ζητήματα. Όλε αυτέ τι γεμμένες περιπτώσεις πάντως, σε γιατί που αναφέρατε θα τις εξετάσω με προσοχή. Μπελία, για τους πράσινους. Κύριε Επίτροπε. Και εγώ θα ήθελα να σα πω κάτι για την ε, βιοποικιλότητα πάρα πολύ χαιρετίζουμε το ότι τα προβλήματα εκεί πέρα τα λαμβάνεται ως υπόψη ως προτεραιότητα και για τους νέους στόχους της Ευρώπης με νέο όραμα, ούτως ώστε να προχωρήσουμε έτσι προς το 2010. Οπότε χρειάζεται πολιτική δέσμευση, χρειάζεται καινούργια πρόθεση του στόχου αυτή για την προστασία επικοινωνία και ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν, κυρίως σε σχέση με τι έγινε στην Κοπενχάγη, και άρα ε, έτσι να αργήσουμε και για την αλλαγή στο κλίμα. Έχω τρεις ερωτήσεις στα πλαίσια αυτής της θέσης. Εσείς θεωρείτε ότι δεσμεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη βιοποικιλότητα για να ανάληψη δράση και πέραν των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα μέσα δεσμεύεστε ότι θα εξασφαλίσετε την τήρηση της νομοθεσίας του Natura 2000 για όλα τα κράτη-μέλη και ότι δεν θα ε, συρρυκνώσετε την εμβέλεια τη υπάρχουσα νομοθεσίας και τρίτον εσείς θα υποστηρίξετε στα πλαίσια του Κολεγίου των Επιτρόπων μια τέτοια πολιτική που θα διέπει όλες τις ε, επιμέρους πολιτικές. Οικονομική, χρηματοδότηση, γεωργία. Σας έκοψε πολλές φορές ο πρόεδρος, αλλά κατάλαβα τι θέλετε να πείτε, λέει ο κ. Ποτότσνικ, και νομίζω ότι σας έχω εξηγήσει ήδη πώς βλέπω τα πράγματα όσον αφορά το τι θα γίνει με την βιοποικιλότητα. Θα πρέπει να γίνει λοιπόν σε παγκόσμια κλίμακα και θα πρέπει πάντοτε να κοιτάμε τι γίνεται και έξω από την Ευρώπη. Συγκεκριμένο παράδειγμα είναι το τι γίνεται με την παράνομη λιλοτόμηση, με τα δάση. Θα πρέπει επομένω να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην βλάψουμε τα ίδια εκείνα και στην Ευρώπη και εκτός αυτής. Άρα σας πω το καταφατικά, έτσι θα πρέπει να δούμε το θέμα παγκόσμια τώρα για το Natura 2000. Νομίζω το είπα προηγουμένως, σαφώς, το τι πρέπει να κάνουμε και από πλευράς διεθνών δεσμεύσεων και των όσων δεσμευόμαστε να κάνουμε. Υπάρχουν δύο τεινά που, κατά τη γνώμη μου, είναι οι βασικές προτεραιότητες. Πρώτον, η συνάντηση της Ναγκόγια περί τα τέλη του 2010 σε σχέση με κάποιου στόχου που θα ασχίσουν παγκόσμια και εκεί θα πρέπει ξεκάθαρα να κατέβουμε για να πούμε ποια είναι η θέση μας. Εκεί θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρες απόψεις και υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο επίσης με ενδιαφέρει πάρα πολύ και αφορά την IPCC, την πολιτική, που θα πρέπει να ισχύσει και για την αλλαγή του κλίματος που είναι ένα παράδειγμα εξαιρετικό για το πώς η γνώση η επιστημονική μπορεί να κατευθύνει τις αποφάσεις των πολιτικών. Δευτερολογία. Αποτελεσματική πολιτική σημαίνει να υπάρχουν παναγία μέσα ελέγχου, εποπτείας αλλά να υπάρχουν και αναγκαίοι πόροι που να αντιστοιχούν στις, στους στόχους. Οπότε σε σχέση με αυτό θα αυξήσετε την αντίστοιχη προοικοδότηση, ας πούμε για το Natura 2000 και στην Κομισιόν και έναν των κρατών μελών θα υποστηρίξετε το να έχουμε υποστήριξη χρηματοδοτική κάποιων ε, προγραμμάτων ε, που θα ωφελούν θα υποστηρίζουν τους φυσικούς πόρους και κάποιο είδου ευαίσθητε τοποθεσίε που θα πρέπει να προστατεύονται. Ποτό είναι ναι, σας απαντώ και η προσέγγιση μου είναι η εξή. Αν ρωτάει κανείς πώς, πώς παραγωγική βοήθεια θα έπρεπε να δοθεί, εγώ θα έλεγα 155 δις και στα πλαίσια της ε, γεωργικής πολιτικής και ε, όσον αφορά τα δικά μου στενά θέματα που δυστυχώς αφορούν ε, πόρα πολύ λίγους πόρους. Άρα, θα πάει στον Αντρό 2000 ένα σημαντικό ποσό και όσον αφορά τις μέλους εξελίξεις θα πρέπει να έχουμε capacity building, δημιουργία δυνατότητα στα κράτη-μέλη και επίσης η προσέγγιση μου χαρακτηρίζεται από το ότι θέλω να είμαι ρεαλιστής. Ξέρω. Ποτέ δεν θα μπορέσω άμεσα να κανονίσω το πόσα χρήματα θα δοθούν σε σχέση με το πόσα πιστεύω ότι χρειάζονται. Αυτό το ξέρουν οι συνάδελφοι. Προθέτω να υπάρχει ένα δίκαιο ποσό το οποίο να δεσμεύεται για αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Τζούλι Γκέρλινγκ. Εγώ θέλω να επανέλθω στην υλοτόμηση την παράνομη. Η αυτή το κόμμα των Τόρις, να θεσπίσει ως νέο έγκλημα την παράνομη υλοτόμηση του Ηνωμένου Βασίλειου. Όμως στην Ευρώπη τίποτα δεν έχει γίνει. Θέλουμε αναμονία. Στη ΣΥΠΑ πρόσφατα αναθεωρήθηκε νομοθεσία ενός αιώνα, ούτω ώστε ό,τι δραστηριότητα έχει σχέση με την παράνομη υλοτόμηση να είναι έγκλημα του ποινικού δικαίου. Αδίκημα του ποινικού δικαίου. Οπότε, δεσμεύεστε εσείς να προσπαθήσετε να έχουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοιου είδους νομοθεσία. Γιατί στο Συμβούλιο δεν τα έχουν βρει ακόμα. Τι λέτε. υπήρξε κάποια κίνηση για εφαρμογή σχετικής νομοθεσίας, κάτι όπως να κάνουμε για την παρανομή υλοτομία. Είχαμε τον Νοέμβριο του 2009 συμφωνία με την Κάνα. Και τώρα θα δούμε αν μπορούμε και με άλλα κράτη να συμφωνήσουμε. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο και οι άλλες χώρες που εξάγουν προς την Ευρώπη εάν θα προχωρήσουν όπως η Γκάνα. Το 2008 θεσπίστηκε κάποια νομοθεσία και τώρα βρίσκεται στη φάση της συναπόφασης. Και υπήρχε μια πόλη στο Συμβούλιο. Μερικοί λέγανε ότι θα πρέπει να έχουμε απαγορευτική προσέγγιση, άλλοι έλεγαν ότι θα πρέπει να έχουμε την πολιτική της επιμελούς διαχείρισης. Και από όσα κατάλαβα πόσα ξέρω. Θα... Το, το κατά πόσο υπάρχει απαγορευτική προσέγγιση θα εξαρτάται από το πόσο εφαρμόσιμα θα είναι, θα είναι τα μέτρα που προτιθέμεθα να πάρουμε γιατί υπάρχουν σημαντικά προβλήματα με την εφαρμογή τέτοια νομοθεσία. Σα υπόσχομαι ότι θα εξετάσω τι λεπτομέρειε του θέματο. Ξέρω Υπάρχει τώρα κάποιο νομοθέτημα με προσέγγιση ε, επιμέλειας μελούς διαχείριση που προωθείται, αλλά θα πρέπει να είμαστε πιο δυναμικοί, πιο ενεργοί στην πολιτική μας και να σταματήσει η, η, καταστροφή των δασών. Και άλλωστε έτσι προκαλούνται για, για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Γκέρλινγκ. Πάρα πολύ χαίρομαι που αυτό θα το λάβετε υπόψη, θα, το, θα σας απασχολήσει και όπως είπα και προηγουμένως θα ήθελα να σας απασχολεί λίγο πιο έντονο αυτό το θέμα πάντως και πάλι καλά Ποτότσνικ. Εάν κάτσετε και δείτε τι έπρεπε να μελετήσω κατά τις διακοπές θα καταλάβετε γιατί όλα αυτά τα θέματα με απασχολούν. Ναι, Ξέρω ότι είναι σοβαρό θέμα και έτσι θα το, χειριστούμε. Υπάρχει κάποιο για τους μη γραμμένους. που θέλει το λόγο, λέει ο πρόεδρος. Η Ελιζαμπέτα Γκαρντίνη. Για να ξαναδούμε λίγο την ε, ε Κοπεχάγη, γιατί ήδη μας απασχόλησε κάπως. Για, για πέστε μου. Ήταν μια αποτυχία. Το βλέπαμε να έρχεται. Δεν θα έπρεπε στα σοβαρά να προβληματιστεί η Ευρώπη όσον αφορά τα μέτρα τα οποία θέλαμε να θεσπίσουμε και είναι τόσο, τόσο, τόσο ε, δύσκολο να εφαρμοστούν παρά το ότι μας απασχόλησαν τόσα χρόνια για να εκπονηθούν. Δηλαδή, έχουμε όλα αυτά τα, τα, τα μέτρα ελέγχου του εμπορίου και δεν καταλήγουμε οι χώρες να θέλουν τον παλιό φόρο του διοξιδίου. Δεν πρέπει η να κάτσει και να προβληματιστεί, να σκεφτεί κατά πόσο θα πρέπει να έχουμε και σταθμιστικά μέτρα στη μεθόριο, στα σύνορα. Δεν θα πρέπει αυτό να μας απασχολήσει. I να σα απαντήσω όσον αφορά την πολιτική πτυχή. Τον σου ρωτήσατε τι θα γίνει μετά την Κοπενχάγη. Ναι, νομίζω ότι ήταν ένα σκληρό μάθημα η Κοπενχάγη. Από μια μεριά έχουμε τους στόχους και τις δεσμεύσεις, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ σοβαρά από πλευράς του Πώς οργανώμαστε εδώ στην Ευρώπη, τι μπορούμε να πετύχουμε, να αλλάξουμε τη δική μας. Και έτσι θα πρέπει να αποκτήσουμε μία φωνή. Να φροντίσουμε να έχουμε περιθώριο λιγμός της διαπραγματεύσεις. Αλλιώς θα μπούμε στο περιθώριο. Και αυτό το προσπαθούμε να κάνουμε και να δεσμευτούμε σχετικά είναι το να γίνουμε τελικά πρωτοπόροι, αλλά δεν τα καταφέρνουμε. Το σημαντικό πάντως στην υπόθεση αυτή είναι το εξή. Γιατί έτσι προχωράει και η έρευνα και η ανάπτυξη όταν ήμουν εγώ εκεί πέρα. Έτσι προχωρούσε. Γιατί α, το θέμα αυτό δεν το παίζουν σοβαρά κάποιοι όπως είπα, αλλά κάνουν λάθος. Για να κάτσει κανείς να δει πόσο χρήματα επενδύουν οι Αμερικανοί. Άρα κακώς πιστεύω ο κόσμος ότι δεν τους απασχολεί. Απλώς οι Αμερικάνοι έχουν τη δική τους, τη δική τους προσέγγιση. Κάνουν το δικό τους, όπως είπε στο τραγούδι του και ο Φρανκ Σινάτρα. My way. Επομένως, να μην υποτιμούμε τα πράγματα, μην υποτιμούμε. Το τι κάνουν, γιατί πολλές φορές αντί να προσέχουμε την ουσία, αναλωνόμαστε στις εντυπώσεις. Eh. Σας ευχαριστώ για αυτή την προσέγγιση. Κάτι ίσω πιο συγκεκριμένο, στρεφόμενοι στι οδηγίε όσον αφορά την ποιότητα του αέρα, γιατί είμαι πεπισμένη ότι δεν ε, εφαρμόζονται πάντα με τον ίδιο τρόπο. Θα ξέρετε πολύ καλά πως υπάρχουν μεγάλες επιφάνειες Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου είναι δύσκολο να υπάρξει η τήρηση των ορίων γιατί ακριβώς υπάρχουν διαφορετικές ε, ιδιαιτερότητες μάλλον γεωγραφικές και κλιματικές και καθιστούν την εφαρμογή αυτών των ε, ορίων πιο δύσκολη. Ας πούμε, εγώ επειδή είμαι Ιταλίδα, είμαι από την Παδανία, 27 ε, εκατομμύρια κόσμος κατοικεί εκεί, έχουμε μια έναν μέσο όρο εκπομπών κάτω από το μέσο όρο, αλλά έχουμε δυσκολία να τηρήσουμε τα όρια. Μπορείτε να σκεφτείτε κάποιες σχετικές ε, διευκολύνσεις για να βοηθήσετε. Είχα ήδη ε, το ίδιο πει προηγουμένως, τώρα υποβάλλετε εσείς με διαφορετική ερώτηση. Ε, θα πρέπει να παραμείνετε στο ίδιο θέμα της ερώτησης και προηγουμένως δεν επέτρεψα την συμπλήρωση. Έχουμε στο τέταρτο γύρο. Η κυρία Κριστίνα Βουτήρα Κουρτίνης έχει το λόγο. Παρακαλώ. Μπράβο σας, γιατί καλά τα πήγατε προηγουμένως. Άλλωστε βλέπετε τα πράγματα ρεαλιστικά. Οπότε πολύ σωστά μα τα λέτε ότι είναι, θα πρέπει να βλέπουμε ολιστικά, σφαιρικά και άρα χρειάζεται συντονισμό, όπω είπατε και με ενδιαφέρει το ότι θα πρέπει τελικά να είμαστε λιγότερο συναισθηματικά φορτισμένοι. Θα πρέπει πιο ε, επιστημονικά να κινούμεθα. Έχουμε ένα σωρό παράπονα διότι ε, και η νομοθεσία και τα έγγραφα που, που παράγεται και που έχετε παράξει στο παρελθόν είναι πιο πολύ συναισθηματικά φορτισμένα και από το αντιμετώπισης παρά επιστημονικής μελέτης. Η Κοπενχάγη θα πρέπει να μας οδηγήσει σε μια τέτοια σφαιρική αντίληψη για την πολιτική που πρέπει να ασκήσουμε. Να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε καλύτερα τι γίνεται με την γεωργία, επί τις εκπομπές και θα πρέπει να δούμε το πώς θα αποκτήσει τα μέσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να έχει το σωστό συντονισμό, να προχωρήσει σε καλύτερη χρηματοδότηση. Δηλαδή θεσμική αντιμετώπιση του, του ρόλου της Κομισιόν και ό,τι δεν έχετε θα πρέπει να το, να το επινοήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ευχαρίστηση ήταν και δική μου στην Η ε, απάντηση θα σας φέρει περίεργη, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε κατά μέρος τα συναισθήματα γιατί είμαστε άνθρωποι. Και τα συναισθήματα είναι ανθρώπινα. Καμιά φορά βέβαια υπάρχει έλλειψη κατανόησης ή και γνώσης ορισμένων πραγμάτων. Where we were certainly one area of the... Ε, ένα τομέα στον οποίο θα πρέπει να εργαστούμε είναι η βελτίωση του επίπεδου γνώσεων για το τομέα. Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, από όσοι θυμάμαι, είναι πολύ πράσινο. Θα πρέπει να εξετάσετε όλες τις πτυχές, όχι μόνο το περιβάλλον, και τις μεταφορές, ενέργεια, νανοτεχνολογία, υλικά, κοινωνικο-οικονομική έρευνα, όλα αυτά θα μπορούσε να πεις ότι το πρόγραμμα πλαίσιο είναι περιβατολογικό και κινείται προς το κατεύθυνση. Όλα τα μέσα που υιοθετήσαμε, τα μέσα που υιοθετήσαμε είναι προς την κατεύθυνση αυτή. ότι θέλαμε δηλαδή να είναι πιο ισχυρή η συνεργασία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για πιο πράσινα προϊόντα, για πιο πράσινη βιομηχανία, για πιο πράσινα σπίτια στα οποία ζούμε. Πάνε έχουμε αυτή την ιδέα κατά Όταν εξετάζουμε τα σημερινά οικονομικά θέματα, είναι ιδανική ευκαιρία να λάβουμε υπόψη μας το όραμα του μέλλοντος προς τα που θέλουμε να κινηθούμε. Σας ευχαριστώ. αλλά εγώ θέλω να επανέλθω στο εξή. Το πρόβλημα του συντονισμού είναι, είναι κάτι το οποίο πρέπει να αφορά ούτε τον Επίτροπο, τον Αρμόδιο, το σύνολο της Κομισιόν, αλλά είναι θέμα δεύτερου, τρίτου επίπεδου διοίκηση. Τώρα με ακούτε? Α, ωραία. Σας τα ξαναλέω σε δεύτερο τρίτο επίπεδο στη δίκη θα πρέπει να αυτό το οποίο είπαμε. Αυτό το οποίο με απασχολεί είναι οι εμπλεκόμενοι οι οποίοι πάντοτε στην Επιτροπή του Περιβάλλοντος επηρεάζουν πολύ τα πράγματα. Η πολιτική της προσαρμογή στο κλίμα, η πολιτική των διευθυντικών ταμείων απαιτούν μεγαλύτερη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης ή της περιφερειακής διοίκησης ε, να επηρεάζουν αυτοί περισσότερο και όχι τόσο πολύ οι εμπλεκόμενοι υπόλοιποι. Συμφωνώ το με αυτό το οποίο είπατε. Συμφωνώ απόλυτα. Ε, έχουμε το πρώτο επίπεδο συνορισμού, αλλά βέβαια δεν αρκεί. Ο ρόλος σας εδώ θα πρέπει να είναι ισχυρό. είναι σαφές αυτός, αλλά όταν αφάνω, αναφερόμαστε για τις επιτόπου πολιτικές, έχουμε σημαντικά μέσα που χρησιμοποιούμε και αρκετά σωστά ήδη. Και είναι καλή αυτή η στιγμή στην οποία ζούμε, γιατί θα δούμε πώς θα έχουμε τις μελλοντικές ε, δημοσιονομικές προβλέψεις. Και αυτά τα θέματα πώς θα εξετάσουμε όλα τα προβλήματα μέσω των προτεραιοτήτων των πολιτικών θα πρέπει να είναι πάρα πολύ έντονο στο μυαλό μας όταν συζητάμε τα θέματα των δημοσιονομικών προβλέψεων. Γεωργία, έχουμε 7% εργαζόμενους από το του πληθυσμού και αυτοί ασχολούνται με το 5% των γιών. Μπορούμε να τους παραβλέψουμε. Είναι η κυπουρή μας αν θέλετε. Ας Βέσλον, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ για τις απαντήσεις που δώσατε για το Rich. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να ενδυναμώσετε την νομοθεσία για τι χημικέ ουσίε, ιδίω για τι χημικέ ουσίε μικρών ποσοτήτων που δεν καλύπτονται από το ρίτσο αυτή τη στιγμή. Θα απαντήσω εδώ μόνο επί της αρχή δυστυχώς δεν γνώριζα τις λεπτομέρειες. Το ρίτσο πάει αρκετά μακριά. και ορισμένα θέματα σχετίζονται και με τις διεθνείς μας συμφωνίες. Αν υπάρχουν λοιπόν θέματα που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, θα εξαιτήσω εις βάθος, βασιζόμενοι στα δεδομένα και αν χρειαστεί μετά να υποβάλουμε προτάσεις για νέα μέτρα, οπωσδήποτε δεν θα διστάσω να το κάνω. Δεν θα θέλουν να κινηθούν προ την κατεύθυνση αυτή. Ένα από τα πολύ επικαιρά θέματα είναι το θέμα της νανοτεχνολογίας, Φερρυπίν. Χωρίς να αναλαμβάνω καμία δέσμη αυτή τη στιγμή, είναι όσο πάει και πιο προφανές ότι η νομοθεσία ρήψη δεν είναι επαρκής. και πρέπει να καταλάβουμε τα θέματα πολύ καλύτερα. Παραδείγματος στο τομέα της ναύνοαυτοκλήχειας που οικονομικά προ... προσφέρει πολλά. Τουλάχιστον υπόσχεται πολλά να προσφέρει. και δεν έχει κανένα συμφέρον. Οπωσδήποτε όχι η βιομηχανία, ούτε εμεί που θέλουμε ασφαλή προϊόντα και σωστά προστατευόμενα. Αυτή η λογική θα πρέπει να ακολουθεί. Γιατί εν τελευταία αναλύση αυτό αφορά όλους που θέλουν να εργαστούν και στο μέλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν η κοινή γνώμη δεν είναι στο μέρος μας βέβαια δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ευχαριστώ, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας για την τεχνολογία. Θέλω να είμαι πιο συγκεκριμένη όσον αφορά τις χημικές ουσίες. γιατί σήμερα τα μωρά στο, στην Ευρώπη εκτίθενται, σε διάφορες ουσίες που είναι στις πλαστικές μπουκάλες γάλακτος παρόλο που δεν μπορούσαν να έχουν πιο ασφαλή μέσα. Κοιτάξτε, εγώ δεν γνωρίζω την υπόθεση αυτή τη λεπτομέρειες. Δεν μπορώ να πω ούτε ναι, ούτε όχι, ούτε τίποτα. Μπορώ να σα υποσχεθώ ότι θα εξετάσω τι λεπτομέρειε. Εάν συζητάμε για επικίνδυνε ουσίε, αν μιλάμε για ουσίε με αρνητικές επιπτώσει, αν αυτό είναι ένα δεδομένο που αποδεικνύεται επιστημονικά, δεν μπορούμε παρά να δράσουμε. ευχαριστώ πολύ. Μάρατ Μακίνες. Ελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε ε, ε Επίτροπε, θέλω να επιμείνω και εγώ σε αυτό το θέμα του ρίτσου και ε, φαντάζομαι θα λάβετε υπόψη ότι και επισκεφτείτε τη σχετική υπηρεσία στη Βιλανδία. Η υπηρεσία αυτή είπε ότι αυτό το έτος θα είναι το πιο προκλητικό και έχουν διάφορε διάφορες υποθεσμίες που πρέπει να τηρήσουν. Πιστεύουν, πιστεύετε ότι η υπηρεσία έχει επαρκείς πόρους για να πληρεί τι απαιτήσει ιδίω όσον αφορά την εφαρμογή τη νομοθεσία REACH, όσον αφορά κυρίω την εφαρμογή τη τιμή έψιλον και πώς θα εξασφαλίσετε να μπορέσουν να ληφθούν υπόψη και οι ανησυχίες βιομηχανίας και όχι μόνο να τηρηθούν οι στόχοι του ΡΙΤΣ και ίσως να χρειαστεί παράταση κάποιων προθεσμιών. Όπως είπα, για, οι διαπρομές για το ΡΙΤΣ ήταν μακροχρόνιες και δύσκολες. Και τώρα φτάνουμε σε μία νομοθεσία που υπάρχει και η κύρια μας ανησυχία είναι να την εφαρμόσουμε. Μία από τις ανησυχίες είναι αυτή που τονίσατε. Υπάρχει το πρόβλημα του ανθρώπινου δυναμικού και όχι μόνο στην υπηρεσία του Ελσίνκη. αλλά και στους άλλους που πρέπει να την εφαρμόσουν στη βιομηχανία και στην Κομισιόν την ίδια. Εγώ βρήκα ότι κάνω τεράστιες προσπάθειες. Δεν θα πρέπει νομίζω να υπερτιμήσουμε. Εγώ καθίδησα κατά τη διάρκεια της εντολής μου δύο ε, διακανονιστικές υπηρεσίες και έμαθα ότι κάθε υπηρεσία χρειάζεται χρόνο πριν να μπορέσει να λειτουργήσει πλήρως. και δεν είναι εύκολο σε ένα-δύο χρόνια να υπάρξει μια νέα οργάνωση και να περιμένουμε όλα τα άλλα ε, που έχουν εξελιχθεί εντωμεταξύ θα μπορούν να εφαρμοστούν, να από την πρώτη στιγμή. Ε, δεν ξέρω τι προβλήματα έχουν με προσωπικό αλλά η ευθύνη δική μου μαζί με τον συνάδελφο Τεζάνη είναι να υπάρχει το επαρκές δυναμικό για να μπορέσει η εφαρμογή να είναι μια πραγματικότητα. <clears throat> Από ό,τι καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή, αυτό είναι ένα θέμα έντονης ενσυχίας. Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να για παρατάσεις. Είναι πολύ νωρί νομίζω. Δεν θα είναι τόσο στο μήνυμα αυτή τη στιγμή να απευθύνουμε. Σημαντική ερώτηση. Δεν μπορείτε να σχολιάσετε ότι αν χρειαστεί κάτι τέτοιο θα γίνει. Γιατί απαντήσατε μεν μακροσκελώς, αλλά όχι σαφώς. Αν υπάρχουν πότε τέτοια προβλήματα θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν. Επίσης το θέμα ήταν κατά πόσον ορισμένες από του ΡΑΣ θα ενταχθούν στο ΡΙΤΣ. Ορισμένε βιομηχανικέ μονάδες έχουν ανησυχίε. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να γίνει ή ίσως δεν γίνει άμεσα. Δεν έχω άποψη. Ξέρω τα πράγματα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, είναι, έχουν υψηλή προτεραιότητα στην ε, ατζέντα μου. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να αναλάβω μια υποχρέωση ότι θα κάνω αυτό τώρα και θα κάνω εκείνο πιο αργότερα. Ξέρω ότι τα θέματα είναι επίγοντα, ξέρω ότι θα γίνουν, αλλά δεν μπορώ να πω παραπάνω και εκτός αυτού δεν είναι μόνο δική μου ε, ευθύνη. Πρέπει να συζητήσω και με τους ε, συναρμόδιους συναδέλφος. Μπορώ να σας υποθέσω, θα εξετάσω το θέμα προσεκτικά και θα δράσουμε. Πρώτα σε ευχαριστώ. Ιούστος Παλέτσκης. Ευχαριστώ. Για να μπορέσει κανένας να ζει φιλικά προς το περιβάλλον, καλό είναι, τίμιο, ευχάριστο, αλλά δεν συμφωνούν όλοι το, ο τρόπος ζωής εξαρτάται και ποια θα είναι τα οικονομικά κίνητρα που θα προτείνετε εσείς για να προωθήσετε φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο ζωής. Να μην υπάρχει σπατάλη φυσικών πόρων, παραδείγματος χάρη. ούτω ώστε να μπορέσουν να υπάρχουν κάποια μέσα για να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Ναι, πολύ σύντομη απάντηση. Ναι. Γιατί πιστεύω ότι πρέπει να αρχίσουμε την αρχή. Και αν ε, το κόστος είναι μέσα στο κάθε προϊόν, θα πληρώνει ο καταναλωτής το πραγματικό κόστος. παραμένει πάλι, αν θεωρήσουμε ότι θα πρέπει να έχουμε μια ανηφόρο μελλοντική ε, κοινωνία και χαμηλή τιμή ενέργειας, ονειροπολούμε απλώς. Δεν είναι αυτό αληθινό. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας όλες τις πτυχές. Ζούμε σε μια οικονομία της αγοράς και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι και αυτό είναι ένα τμήμα του σκεπτικού μας. Και θα πρέπει να το Αυτό που είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουμε είναι να έχουμε από τη μια μεριά την αεφορία και από την άλλη μεριά την αύξηση του ΑΕΠ. Θα πρέπει λοιπόν να βασιστούμε στην, ε, και στα δύο. Να χρησιμοποιούμε λιγότερους πόρους Εύκολο να το πούμε, δύσκολο να το πραγματοποιήσουμε. Μια από τι ιδέε που θα ήθελα να ακολουθήσω είναι αυτή εδώ που σα δείχνω. Η ιδέα τη διαχείριση των πόρων. Έχουμε το προϊόν στο μέσον. Έχουμε πολύ συγκεκριμένη νομοθεσία όσον αφορά τα, τα απόβλητα, αλλά το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι το καλύτερο απόβλητο είναι το μη απόβλητο, να μην υπάρχει δηλαδή απόβλητο. Θα πρέπει λοιπόν να συγκεντρωθούμε στα πρώτα δύο τμήματα. Παραγωγή και κατανάλωση. Πώς παράγουμε. Και υπάρχουν πολλά εδώ. Από την οδηγία οικολογικής αποτελεσματικότητας, ε, οι δημόσιες αγορές, ε, ε, ε, που να λένε ότι κάποιο προϊόν είναι φιλιτό. Όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ για τις πιστικές σας απαντήσεις, Πρόεδρε. Μετά από δύο ώρες όλοι έχουμε κάπως κουραστεί, ιδίως εσύ. Αλλά ειλικρινά, στην αρχή της ακρόσης νόμιζα ότι είμαι στο θέατρο. Άκουσα χειροκροτήματα. Πότε δεν έχω ξανακούσει τόσα πολλά χειροκροτήματα σε τέτοιε ευκαιρίες. Ούτε τώρα, ούτε πριν από πέντε χρόνια. Συγχαρητήρια λοιπόν. Και έχω μια πολύ προσωπική ερώτηση. Στην καθημερινή σας ζωή τι κάνετε για να διασώσετε τον πλανήτη μας. Yeah, first, uh, first comment about the I would prefer it... Καταρχήν, Πραγματικά θα προτιμούσα το χειροκρότημα να έρθει μετά από πέντε χρόνια και όχι σήμερα. Αλλά και το σημερινό καλό ήταν, δεν λέω. Ε, τώρα, τι κάνω καθημερινά. Προσπαθώ να σκέφτομαι ως υπεύθυνο πολίτης. Τώρα ρωτάτε αν, ε, αν ε, χωρίζω τα δικά μου σκουπίδια, ναι, τα χωρίζω. Σε διαφορετικούς σκουπιδοντενικέδες. Τώρα, άμα ρωτάτε τι αυτοκίνητο οδηγώ, μάλιστα μπορούμε εύκολα να συγκρίνουμε τις σημειώσεις με τον προκάτοχό μου, γιατί ήμουν ε, ιδιοκτήτης ε, του Price στο σπίτι μου ε, το 2004, όταν ακόμα ήταν το πρώτο που είχε βγει στην αγορά. Να σας πω ότι λειτουργεί εξαιρετικά καλά. Να σα πω, το τέλο τη ιστορία στα πέντε λεφτά, καθώ τα κλείνω. Γιατί η... ιστορία δεν έχει τόσο happy end. Ναι, προσπαθώ λοιπόν ό,τι κάνω να ε, ται, ταιριάζει. Γενική ερώτηση λοιπόν με αυτή την επερώτηση, αλλά έχουμε κάποια επιπλέον στοιχεία. Συζητού, συνεχίζουμε με τον Σαλβατόρη Ταταρίλα. Κανένα δεν έχει κουραστεί γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα τα όσα ακούμε. Είναι... Είμαστε φρέσκοι φρέσκοι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, ο στόχος να περιοριστεί η παγκόσμια θέρμανση του πλανήτη εντός των δύο βαθμών Κελσίου στοχεύει στο να αντιστραφούν οι αρνητικές συνέπειες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον που περιλαμβάνουν και την απώλεια της βιοποικιλότητας και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος αλλά και τη διατήρηση του αέρα, του νερού, των δασών κτλ. με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Όλα αυτά είναι ε, κίνητρα τα οποία συμμεριζόμαστε. Όμως υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που αποδεικνύουν, ότι, που μάλλον που θεωρούν ότι ο στόχος των δύο βαθμών είναι ανέφικτο Πρακτικά, ορισμένοι επιστήμονες μιλάνε για την ε, μεγάλη αυταπάτη των δύο την ψευδέστηση των δύο βαθμών. Εσάς ποια είναι η αποψή σας σε σχέση με αυτό το πρόβλημα και ιδιαίτερα ποιος είναι ο δικός σας ρόλος, η θέση σας ως Επίτροπος Περιβάλλοντος, πώς τοποθετήσετε ενώπιον μιας πιθανής αύξησης του στόχου από τους δύο στους τρεις βαθμούς Κελσίου. Ευχαριστώ. Πρώτον, ελπίζω να επαναλάβετε την ερώτηση στον συνάδελφό μου σε δύο μέρες. Ελπίζω να μην περιμένετε από τον ε, ενεργό ακόμη Επίτροπο Έρευνας και Ανάπτυξης να σας πει τίποτα άλλο εκτός από το ότι θα παραμείνουμε στο επίπεδο που η επιστήμη έχει προβλέψει. Εμείς προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας καθημερινά. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε ακόμα και μπορώ να σας επαναλάβω ότι είμαστε ευτυχείς που έχουμε το Διεθνές Πάνελ για τι κλιματικέ αλλαγέ που έχει κάνει εξαίρετη δουλειά. Έχει κάνει εξαίρετη δουλειά γιατί όχι μόνο γιατί οι μεγαλύτεροι επιστήμονες, σπουδαίτεροι επιστήμονε είναι συγκεντρωμένοι εκεί, αλλά γιατί έχει βελτιωθεί η γνώση του κοινού, το, του ευρέω κοινού, ότι πραγματικά παίρνουμε σοβαρά το θέμα. Πάντοτε υπάρχουν στιγμές δυσπιστία ή μεγάλη εμπιστοσύνη, αλλά έτσι, έτσι λειτουργεί και η επιστήμη. Είναι πολύ καλό που υπάρχει ένα σώμα που εσείς, εμείς ως υπεύθυνοι για τη λήψη των πολιτικών αποφάσεων να μπορούμε να βασιστούμε και να έχουμε τη δυνατότητα να βασιστούμε σε κάτι το χειροπιαστό. Θα θυμάστε ότι ο πρόεδρος Μπαρός υποσχέθηκε πως θα έχει έναν ε, ε, παριθμόν ένα επιστημονικό σύμβουλο στο σώμα της Κομισιόν. Πολύ σημαντική πρόοδος και αυτή, αλλά αν είναι 2 ή 3% τώρα. Η απάντησή μου είναι, δεν ξέρω. Ελπίζω να είναι το δύο, οι δύο βαθμοί ε, εφικτοί και να μπορέσουμε αρκετά σύντομα να λάβουμε και τα απαραίτητα μέτρα. Αλλά ούτω ή άλλω, είτε με το 2 ή με το 3%, του 2 ή του 3 βαθμού, θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Θα πρέπει ήδη να λάβουμε τα απαραίτητα προσαρμοστικά μέτρα. Ναι, θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Ωστόσο πιστεύω ότι για να επιτύχουμε το αποτέλεσμα αυτό θα πρέπει να υπάρξει ρίζη κρυξικέλευθη αλλαγή στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, σας ρωτώ, είναι καλή η πολιτική να υποδεικνύουμε από τη μια πλευρά περιβαλλοντικούς στόχους που δεν είναι εφικτοί ρεαλιστικά και απ' την άλλη να μην κάνουμε τίποτα για να συγκεντρώσουμε, μάλλον να θεσπίσουμε μέτρα που θα μπορέσουν να αλλάξουν τη δική μας, ε, τον τρόπο ανεφοδιασμού σε ενέργεια. Concerning the... The energy, uh, my answer would... Σε σχέση με την ενέργεια, η απάντησή μου είναι πως θα συμβεί. Το θέμα είναι αν θα γίνει αρκετά σύντομα. Θα συμβεί. Αυτό σας το εγγυώμαι. Σε 50 χρόνια πρόβλεψή μου είναι ότι τα οι μεγαλύτερες ενεργειακές δυνάμεις στον κόσμο δεν θα είναι αυτές που θα έχουν το πετρέλαιο, αλλά αυτές που θα έχουν την πιο προηγμένη τεχνολογία που θα είναι περιβαλλοντικά φιλική. Νομίζω πως προς αυτή την κατεύθυνση οδεύουμε. Τώρα αν προχωράμε αρκετά γρήγορα, αυτό είναι ένα πραγματικό ερώτημα. Αυτό είναι που πρέπει να απαντήσουμε. Και σε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση που ίσως συνδέεται, αλλά δεν θα έχω χρόνο να σας το εξηγήσω, ε, συνδέεται με τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε, για παράδειγμα, στις μεταφορές, δηλαδή μηχανή καύσης. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι εναλλακτικέ λύσεις, να δούμε τις μακροπρόθεσμα βιώσιμες λύσεις. Ε, με αυτόν τον τρόπο νομίζω πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα και είμαι πεπισμένος ότι θα γίνουν όλα αυτά, αλλά ο χρόνος βέβαια είναι καθοριστικό στοιχείο. Next question, Nessa Childers. Επόμενη ερώτηση, Nessa Childers. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε. Θα επανέλθω στην επιβολή ίσως με περισσότερες λεπτομέρειες. Όπως γνωρίζετε υπάρχει μακρά ιστορία ορισμένων ε, κυβερνήσεων που ε, αντιστέκονται ή και παραβιάζουν την περιβαλλοντική νομοθεσία. Έχω λοιπόν δύο ερωτήσεις εδώ. Θέλω να γνωρίζω ποια οι νέοι μηχανισμοί επιβολής θα χρησιμοποιηθούν κατά των εθνικών κυβερνήσεων που συνεχίζουν να παραβιάζουν την περιβαλλοντική νομοθεσία και θα εφαρμόσετε την οδηγία EIA για να θα την προσαρμόσετε μάλλον ώστε να είναι πιο αποτελεσματική στην επιβολή της γιατί είναι ιδιαίτερα προβληματική. Και έπειτα, πώς ε, θα μπορέσετε να αντιπαρέλθετε τους ισχυρισμούς που χρησιμοποιούν την οικονομική κρίση ως δικαιολογία για να μην εφαρμόσουν επαρκώς την περιβαλλοντική νομοθεσία. Ε, κοιτάξτε, ένα, κάτι το οποίο προσπαθούμε να λύσουμε και που ετοιμάζουμε είναι ότι έχουμε πολλά, βέβαια πολλά παράπονα, πολλές ε, καταγγελίες και βέβαια καταγράφονται και ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία είναι η ανάπτυξη του νέου συστήματος ε, καταγραφής των καταγγελιών. Ε, ε είτε μας αρέσει είτε όχι, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι πραγματικές δυνατότητες για την εφαρμογή και για τον έλεγχο ε, εξαρτώνται από τα κράτη-μέλη. Αυτά δηλαδή είναι στα χέρια των κρατών μελών. Ε, πρόσβαση στην δικαιοσύνη όπου νομίζω πρέπει να συνεχίσουμε με τα τμήματα εκείνα που αποτελούν την ε, ε, νομοθεσία. Με πολλά από αυτά προτίθεμαι να επιμείνω γιατί είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η συνεργασία ανάμεσα σε εμά και τα κρατημέλη. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που θα μπορούσε κανείς να αναφέρει, αλλά σίγουρα ένα αφορά τις επιθεωρήσεις ε, για παράδειγμα, θυμάμαι ότι είχατε το 2007 ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου για το αν χρειάζεται οδηγία ή αν χρειάζεται μια επιθεώρηση των ευρωπαϊκών επενδύσεων. Φέτος το Μάρτιο θα ε, έρθει για συζήτηση και επί τη βάση όλων αυτών θα αποφασίσουμε. Αν υπάρχουν σαφείς, ε, σαφή μηνύματα ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο θα προχωρήσουμε προς αυτή την κατένθεση βεβαίως. Έπειτα, για το EIA είναι μια οδηγία, αν κατάλαβα καλά, που κλείνει το, ε, αργυ... τα αργυρά της γενέθλια, δηλαδή την αργυρή της επέτειο, 25 χρόνια δηλαδή. Εδώ σκοπεύουμε να κάνουμε διαβούλευση και θα έχουμε τη δυνατότητα, θα έχετε τη δυνατότητα να εκφράσετε τις απόψεις για το πού θα πρέπει να, πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε. Και τέλος, στο επόμενο λεπτό θα συνεχίσω. Σας ευχαριστώ. Με καθησυχάζετε με την απάντησή σας και θα ήθελα απλά να ρωτήσω σε συνέχεια της ίδιες ερωτήσεις Με τα θέματα της ε, συμμόρφωσης θα συμμετέχει εδώ το Κοινοβούλιο όσο γίνεται περισσότερο και στο λόγο σε όλο σας το χαρτοφυλάκι. Ναι, βεβαίως. Η, ερώ... απάντηση είναι όσο γίνεται περισσότερο. Εδώ μ, έχουμε αναπτύξει συνεργασία και θα πρέπει να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι πεποίθησή μου ότι έχουμε πολύ ξεκάθαρα ευρωπαϊκά συμφέροντα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ε, ως προς αυτό το θέμα και σίγουρα θα έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. και όθηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Ναι, λοιπόν, η απάντησή μου είναι αυτή και έρχομαι στο θέμα των της οικονομίας που ρωτήσατε ως τέταρτο σκέλος της πρώτης σας ερώτησης νομίζω ότι είναι λάθος αυτή η φιλοσοφία Οποιοςδήποτε δηλαδή δεν κατανοεί ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, έχει λάθο. Η οικονομική κρίση είναι η καλύτερη ευκαιρία για ορισμένε από τι διαρθωτικές αλλαγέ που κανονικά δεν κάνει κανεί αν δεν είναι υποπίεση. Αυτή τη στιγμή είμαστε υποπίεση. Α το χρησιμοποιήσουμε και α προβούμε σε απαραίτητε αλλαγέ. Και πολλέ εταιρείε το καταλαβαίνουν αυτό. Πολλέ κάνουν τεράστιε επενδύσει, τεράστιε καινοτομίε και νομίζω πως αξίζουν σε ξεκάθαρα θετικά μηνύματα και υποστήριξη από την πλευρά μας. Um, uh, Σα ευχαριστώ. Ρωμάνα Γιόρνταν Σίσελ. Και επίτροπε, κερδίσατε ένα καφέ. Πήρα και εγώ έναν για να σας κάνω παρέα. Μια ερώτηση. Επίτροπε, για την ανάπτυξη του προγράμματος Life Plus που χρηματοδοτεί τις καλύτερες πρωτοβουλίες ή τα καλύτερα πιλωτικά προγράμματα για το Natura 2000, του Natura 2000. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όρισε το ποσοστό κατανομής ε, των προγραμμάτων ισόρροπα για τις αναπτυσσόμενες χώρες και τα, κονδύλια έπειτα φτάνουν ε, από τη στιγμή που υπάρχουν συγκεκριμένοι πόντοι για τα συγκεκριμένα προγράμματα. Το 2008 έγινε μια καθόλου ισορροπημένη κατανομή των πόρων και της χρηματοδότησης και αυτή είναι η ερώτησή μου πώς θα ε, μπορέσουμε να κατανείμουμε πιο σωστά και πιο ισόρροπα τα κονδύλια του Life Plus ανάμεσα στα κράτη-μέλη και πώς θα εγγυηθείτε τον έλεγχο των δαπανών και τις ε, δαπάνες μάλλον αυτών των κονδυλίων στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ισορροπία στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Α, ωραία είναι το καφέ. Και έπειτα ωραία είναι να ακούει κανείς και τη γλώσσα του. Το LIFE είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το μεγαλύτερο τμήμα των, κονδυλίων για τα προγράμματα live μέχρι στιγμής ε, είχαν ε, ε, κατανεμηθεί έτσι ώστε να δημιουργηθούν κάποια πάρκα προστατευόμενα μέσα στο πλαίσιο του Natura 2000 και μέσω της οδηγίας για τα πτηνά και τους οικοτόπους. Νομίζω πως ε, θα μπορέσουμε να, έτσι να δημιουργήσουμε ένα χώρο ώστε τα κονδύλια αυτά να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη όλων αυτών των στόχων αλλά και διαφόρων παρεμφερών όπως ε, η ενίσχυση των ε, δυνατοτήτων των κρατών μελών. Όταν ε, ασχοληθήκαμε με τη δαπάνη των ταμείων πιο ισορροπημένα, με ρωτήσατε ποια ήταν η ισορροπία στις δαπάνες αυτές. Δεν ξέρω ακριβώς όλα με λεπτομέρειες όλα τα στοιχεία. Θα πρέπει να δω τα στοιχεία για την κατανομή των κονδυλίων. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα προσέξω πολύ το συγκεκριμένο σημείο και το μόνο που θέλω να υπογραμμίσω άλλη μια φορά είναι ότι τα κονδύλια αυτά είναι πολύ σημαντικά και είναι δίκαιο για με τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές να ενισχυθούν οι στόχοι που έχουμε ενώπιόν μας για το Natura δεν θα πρέπει να αξιολογηθούν μόνο από αυτή την οπτική. Θα είναι σημαντικό να έχουμε μια οριζόντια προσέγγιση και να περιλαμβάνουμε εκεί όλες τις περιβαλλοντικές προτεραιότητες σε όλες τις πολιτικές, στη διαρθωτική, στη γεωργική, σε όλες τις πολιτικές που έχουν επίπτωση, αντίκτυπο μάλλον στο περιβάλλον και στην ερευνητική πολιτική για παράδειγμα και οι πολιτικές εκείνες που είναι πολιτικές κλειδιά και που μπορούν να επιφέρουν αλλαγές. να ε, χρησιμοποιηθούν. Συμφωνώ με την σημασία της οριζόντιας προσέγγισης, όπως είπατε. Και καθώς δεν έχετε στοιχεία, θα πρέπει να σας πω ότι το μεγαλύτερο τα περισσότερα μάλλον κράτη δεν ε, λαμβάνουν ε, χρηματοδότηση, μόνο 9 χρηματοδότησαν το 50% των, ε, της χρηματοδότησης. Αυτό δείχνει το πόσο σοβαρό είναι το θέμα των δαπανών αυτών και θα ήθελα να ακούσω από εσά ότι προσωπικά θα δεσμευτείτε ώστε να αναλυθούν από την Κομισιόν τα αίτια για αυτή την κατάσταση και να υιοθετηθούν κατάλληλα μέτρα ώστε να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Κοιτάξτε, ναι, ξέρω πως υπάρχουν προβλήματα ε, στην χρήση αυτών των ταμείων και των κονδυλίων. Τα όσα είπατε θα το ελέγξω, θα ακολουθήσω την ε, σύστασή σας και θα ασχοληθώ προσωπικά ώστε να γίνει ανάλυση του είδους που λέτε. δεν υπάρχει ήδη, αν δεν υπάρχει ήδη θα την κάνουμε και προσωπικά θα διαβάσω και τα αποτελέσματα για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε τον καλύτερο τρόπο. Σας ευχαριστώ, ο Τόμας Ούλμερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Μαξίφια Επίτροπε, έχω μια ερώτηση που αφορά κυρίως το τεχνικό τομέα συνεργασίας με το Κοινοβούλιο και όχι από τη ουσία θα μπορούσατε να φανταστείτε να δώσουμε προτεραιότητα στα θέματα του περιβάλλοντος όσον αφορά την αποτελεσματικότητα χρήση των πόρων προ θέματα υγείας κλπ. Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσατε να θεωρήσετε ότι θα είχε πιο στην ηγεσία. Και πώς θα φροντίσετε να μην επαναλαμβάνετε η παρουσίαση διαφόρων φακέλων που έχουμε ήδη απορρίψει κάτω από διαφορετική ε, μορφή. Ποια είναι η άποψή σα για τι λεγόμενε sunset clauses ε, της Τρίτη ηλεκτροδοτήρωσης και εκτο αυτού ποια είναι η άποψή σα για στρατηγική για το Δούναβι. I Δεν μπορώ να σας απαντήσω με ακρίβεια τώρα, αλλά σας υπόσχομαι. Πώς? Όλα τα θέματα για το οποίο συνεργαζόμαστε δηλαδή για τα πάντα, ότι όλα αυτά θα τα μελετήσω με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα. Με πάντα αυτή η φιλοσοφία με εμπνέει. Βεβαίω και αυτή η διαδικασία που είπαμε, είναι διαμαρτυρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εμένα με βρίσκει σύμφωνο και η συνεργασία μαζί σα. νομίζω ότι είναι κάτι θετικό, ε, είναι κάτι σημαντικό ότι μπορείτε να επηρεάσετε περισσότερο τώρα τι λήψει αποφάσεων και τελικά από κοινού θα πετυχαίνουμε καλύτερε ε, επιδόσεις Αυτά έχω να σας απαντήσω. Για όλα τα συγκεκριμένα θέματα που μου αναφέρατε δεν έχω τώρα κάποια σαφή εικόνα. Όμως είμαι ανοιχτό, είμαι έτοιμος να σας ακούσω για οποιοδήποτε πρόβλημα. Νομοθεσία και οδηγία ήταν ε, λέξεις που τις είχα ακούσει λιγότερο πέντε χρόνια ή περισσότερο τις άκουσα τώρα εδώ στο κοινοβούλιο στις ακροάσεις. Άλλωστε έχουμε και τώρα και την καινούργια επιτροπολογία. Που νομίζω θα μας δώσει ευκαιρία να συνεργαστούμε περισσότερο. Εμεί ευχαριστούμε ο πρώτος και τώρα πάμε στον πέμπτο και τελευταίο γύρο ερωταπαντήσεων και έχουμε έξι ερωτήσεις. Πρώτος ο Ιωζουά Φεραίρα από την ενωτική αριστερά. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε. Μια από μόνο ένα λεπτό μου αναλογεί σας ρωτώ ευθέως βιοπικιλότητα και συγκεκριμένα χρηματοδότηση της ε, πολιτικής για την βιοπικιλότητα και για το Natura 2000. Συμφωνείτε με το πρότυπο χρηματοδότησης που ισχύει σήμερα προβλέπεται κάτι για το Natura 2000 και εμεί συμφωνούμε σωστά να υπάρχει τέτοιου είδου οριζόντια αντιμετώπιση, εγκάρση αντιμετώπιση. Όμω όμως, πρόκειται για κάποια χρηματοδότηση που προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Γεωργικής Ανάπτυξης ή από τα Διευθυντικά Ταμεία. Συμφωνείτε αυτή η χρηματοδότηση του Natura 2000 να συνεχιστεί ή θέλετε ότι θα πρέπει να ψάξουμε ένα άλλο συγκεκριμένο μοντέλο ειδικό για το Natura 2000. Εσεί είπατε στην επιστολή που μα απευθύνατε ότι θέλετε να υπάρξουν καινούργιοι στόχοι, καινούργιε προκλήσει, καινούργια μέσα πολιτική. Άρα, εσεί βλέπετε να υπάρχει ε, κάποιο πρόβλημα. Και έτσι να μπορέσουμε για τι νέε προκλήσεις να έχουμε καινούργια μέσα πολιτική. Εσεί τι θεωρείτε, ποιο είναι το πρόβλημα, νομίζω ότι είναι πρόβλημα στην πολιτική που ακολουθούμε ή στην, στην χρηματοδότησή της. Όχι, όχι, όχι. Ο Λογικός Επίτροπος για την βιοποικιλότητα ε, κατόπιν των όσων είπαμε σήμερα, δύο μισή ώρες ε, καταλήξαμε, μπορούμε να καταλήξουμε για το ότι έχουμε κάποιες πολύ σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την βιοποικιλότητα, όσον αφορά και την κατανόηση κατάσταση και τη βελτίωσή της. Γιατί πάντα στη ζωή, πάντα για το Natura 2000 Πάντοτε έχουμε κάποια κεφάλαια, ε, κάποιους πόρους και όπως και στη ζωή δεν πρέπει να είμαστε υπεραπλουστευτικοί. Μόνο με μια ολιστική σφαιρική ε, ε, απόκριση, ανταπόκριση, μόνο έτσι μπορούμε να βρούμε κάποιες, κάποιες λύσεις. Από μόνη της η γεωρική πολιτική δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και ε, το ίδιο ισχύει και για, τις, ε, τα αντίστοιχα και κεφάλαια και για την αλληλευτική πολιτική. Και το θέμα τη βιωσιμότητα θα πρέπει μέσα από όλε τι πολιτικέ να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί, εάν έχουμε βιωσιμότητα σε άλλε πολιτικέ, τότε θα βρούμε απαντήσει και για την πολιτική που θα υποστήριξει τη βιοποικιλότητα. Όχι. Δεν λέω τώρα για νέου χρηματοδοτικού μηχανισμού και νέε πολιτικέ, Θα να χρησιμοποιήσουμε ό,τι έχουμε τώρα. Όμω βέβαια θα γίνει κάποια στιγμή συζήτηση για ε, ε, τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές και θα πρέπει να δούμε πώς οι νέες δημοσιονομικές προοπτικές, οι νέες δημοσιονομικές θα βοηθήσουν και την πολιτική για την βιοποικιλότητα. Γκέρλινγκ, για τρίτη φορά. Μάλλον ε, το τώρα πια είχε αποκτήσει ειδίκευση σε αυτό το θέμα. Ή εκτό αν είσαι μόνη που αυτά τα θέματα στην πολιτική σου ομάδα. Είδατε πώ με πιστεύονται, λέει κύριε Γκέρλινγκ. Και έχω μια ερώτηση γενική φύση. Όσον αφορά τον ρόλο σα ευρύτερα στο σώμα των ε, επιτρόπων. Πολλοί από εμά Θεωρούμε ότι η Ευρώπη δεν θα πρέπει να ανακατεύεται με όλα. Αλλά βέβαια δεν πιστεύουμε κάτι τέτοιο για την περιβαλλοντική πολιτική. Επομένως, καλά τα έχει πάει η Ευρώπη, όμως τις χρεώθηκε της Ευρώπης και της Κομισιόν με αποτυχία της Κομεχάγης επομένως. Το θέμα είναι τι συνέπειες θα έχει αυτή η αποτυχία της Κοπενχάγης. Εσείς τι θα κάνει τόσο ώστε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων. Πώς θα μπορείς να ξαναγίνει πρώτα απ' σε αυτά τα θέματα η Ευρώπη όπως ήταν. Επίτροπος, όσον αφορά την Επιτροπή μας, μια που είμαι μέλος της, αλλά μιλώ και για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιστεύω ότι θα πρέπει να προπλησιάσουμε τις προσπαθίες μας. Οι προφάσεις για το κλίμα, οι προφάσεις για το περιβάλλον είναι θέματα ουσίας και επομένως κατά κάποιο τρόπο πολλά θέματα τα οποία δεν ήταν στο επίκεντρο της επικαιρότητα, όπως το νερό, η βιοπικιλότητα. Δεν ήταν στο επίκεντρο της προσοχής, όπως τα απόβλητα και όλα αυτά νομίζω ότι θα ε, είναι αλλιώ το μέλλον. Ακριβώς γιατί τώρα το περιβάλλον θα προσεχτεί περισσότερο. Και αυτό νομίζω ότι είναι θετικό. Τώρα όσον αφορά γενικότερα το ρόλο μας, γενικότερα τις ε, ευθύνε μας. Νομίζω ότι είπα προηγουμένω κάτι σχετικό όταν απαντούσα σε άλλους συνάδελφους. Θα πρέπει να κάτσουμε για να δούμε όλοι πόσο θέλουμε να στρατευτούμε για αυτά τα θέματα, γιατί είναι κάτι που μας αφορά όλους, κάτι το, όπως η αλλαγή του κλίμακος. Επομένως ε, και οι άλλοι τι κάνουν. Να βρούμε κάποια τέτοια προσέγγιση. Άρα, να δούμε πώ η ευρωπαϊκή προσέγγιση που εμεί αναγκαστικά θα έχουμε θα μπορέσουμε να την μεταλαμπαδεύσουμε και στον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί τέτοιου είδου προσέγγιση χρειάζεται όσον αφορά την πρωτοπορία της Ευρώπης, τον ηγετικό τη ρόλο, εάν θέλουμε να είμαστε σοβαροί πολιτικοί, σοβαροί πολίτε, τότε θα πρέπει όντω να αναλάβουμε την ευθύνη μα, εάν πιστεύουμε ότι ισχύουν αυτά τα οποία λέμε. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Είμαστε πρωτοπόροι. Κύριε Επίτροπε, λέει κύριε Χάση, πάρα πολύ σωστά είπατε πρέπει να έχουμε αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Αλλά πέστε μας πιο συγκεκριμένα τι σκοπεύετε να κάνετε. Τι αλλαγές θα επιφέρετε για την επόμενη φοιτεία. Για παράδειγμα, θα τεθούν κάποιοι δεσμευτικοί στόχοι. Και επίσης σε απόλυτα στοιχεία θα βάλετε και επιδημιουργούς στόχους όσον αφορά την μείωση της κατανάλωσης των ενεργειακών πόρων γιατί η αποσύνδεση που έγινε Ε, αφορούσε κάποιες επιδόσεις ε, σχετικές και όχι σε απόλυτα νούμερα. Πρόεδρε, ε, Επίτροπος, πάρα πολύ σημαντικό αυτό που το λέτε και ας έχει βγει μετά από τόση ώρα συζήτηση, γιατί τα πρώτα δύο στοιχεία που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι τα εξή. Πρώτον, ότι η Ευρώπη είναι εισαγωγέας πόρων να δούμε τι κάνουν οι εταίροι μας. Διότι προς ενδιαφέρον το ότι η Ιαπωνία όσον αφορά την αποτελεσματική χρήση των πόρων είναι καλύτερη από εμά. Η μέθοδος της, της ενεργειακής εκμετάλλευσης ΑΕΠ ανατών δεν είναι η πιο καλύτερη μέθοδο Τώρα όσον αφορά ε, το πρόβλημα που θέσατε, ναι, θα είναι στο επίκεντρο της προσοχής μου. Ήδη έχουμε στόχους για την ανακύκλωση. Έχουμε την οδηγία για την, τον ε, οικολογικό σχεδιασμό, βιωσιμότητα, κατανάλωση, την παραγωγή. Υπάρχουν, υπάρχουν όλα τα νομοθετήματα αυτά και επομένως Πρέπει να είμαστε πάντοτε προσεκτικοί για τους στόχους που θέτουμε, για στρεβλώσεις, για μετακύληση του βάρους, του άχθους. Και προσοχή γιατί όλα αυτά είναι περίπλοκα. Όμως θα πρέπει πάντοτε να περιμένουμε όλο ένα και λιγότερο το περιβάλλον. Άρα θα πρέπει να επιβληθεί αποτελεσματική χρήση των πόρων και αντίστοιχη στόχη. Τώρα, να δούμε όχι το πόσα θα ζητήσουμε σαν στόχους, αλλά το πώς θα το πετύχουμε. Αυτό είναι το πιο βασικό και για την αναθεώρηση της θεματικής στρατηγικής και για, τον, για την ανακύκλωση, για διαχείριση των αποβλήτων. Αυτά στο άμεσο μέλλον θα τα συζητήσουμε. Merci, Corinne Lepage. ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, κύριε Υποψήφη Επίτροπε, σα ευχαριστούμε πρώτα πρώτα για τον τρόπο με τον οποίο μα απαντάτε, αλλά εγώ θέλω κάτι άλλο να θίξω το οποίο δεν έχει φύγει ακόμα, δηλαδή όσον αφορά την αξιολόγηση τη εμπειρογνωμοσύνη, κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό για το περιβάλλον. Πώ θα εξασφαλίσετε να υπάρχει τέτοια εμπιστοσύνη από τους ε, πολίτες μας όσον αφορά τις ε, πληροφορίες που τους δίνονται για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Πώς θα βελτιώσετε, πώς θα κάνετε ε, καλύτερη την δήλωση αξιοπιστίας για τη δήλωση συμφερόντων από τους εμπειρογνώμονες γιατί τους χρησιμοποιείτε στην Γενική Διεύθυνση για το περιβάλλον. Μπορείτε κάπως να φέρετε μεγαλύτερη διαφάνεια σε σχέση με τα λόμπι, σε σχέση με την υποχρέωση της ε, εγγραφής τους σε αυτό το μητρό που θέσπισε ο Κάλλας. Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της και να σταματήσει να πιστεύει ότι υπάρχει κάποια αντίφαση στο ρόλο των λόμπι. Ένα, ένα λεπτό. Μόνο μίλησε ο πρόεδρε. Επίτροπος. Πρώτον, να σα ξεκαθαρίσω ότι πιστεύω για τα λόμπι. Νομίζω ότι είναι ένα απόσπαστο τμήμα, φυσικό κομμάτι της δουλειάς μου και παίρνω πληροφορίες από αυτούς και αυτό σημαίνει ότι κάνω ό,τι μου λένε, αλλά πρέπει να ακούω διαφορετικές απόψεις και πιστεύω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να φροντίσω είναι το να ακούω όλες τις απόψεις. Το ίδιο για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δεύτερον, όσον αφορά την ποιότητα των μελετών, κάθε μέρα την προηγούμενη πενταετία ασχολιόμουν με τις σχετικές μελέτες τι έβγαζε η Γενική Διεύθυνση Ερευνών, οπότε ξέρω ότι είναι υψηλής ποιότητας και ότι η διαδικασία της επιλογής γίνεται με τέτοιο τρόπο που είναι αμερόληπτη. Και πολλές φορέ βέβαια μας μπαίνει η αμφιβολία του αν κάτι, υπάρχει κάποια αντίβαση, αν κάτι πάει στραβά. Όχι, αυτό δεν, δεν, δεν έχει καμία θέση στο σύστημά μας. <clears throat> Οπότε αυτά που έκανα και πριν θα τα κάνω και τώρα. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμπιστεύεται κανείς τους εμπειρογνώμονε. Και να εμπιστεύεται κανείς και, αυτά που παράγουν, αυτά που συντάσσουν οι επιστήμονες οι Ήδη έχουμε φέρει κάποιες βελτιώσεις. Και είμαστε κατηγορηματικοί σε αυτό. Στο να έχουμε όσο γίνεται καλύτερη μελέτη των επιπτώσεων ούτως ώστε αυτές οι επιπτώσεων να κάνουν αυτό που πρέπει και να είναι αποτελεσματικές. Τελευταία σημαντική έρωση του κυρίου Ταμπάτζη. Κύριε αυτή η ακρόαση δείχνει σημασία της διαχείρισης του θέματος και θα έλεγα να τελειώσουμε με το θέμα που ξεκινήσαμε, το θέμα της διαχείρισης των υδάτων, γιατί το θέμα των υδάτων είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και για όλο τον κόσμο. Εσείς είπατε ότι σκοπεύετε να συνεχίσετε με την εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα. Για πέστε μας όμως, ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Κανένα από τα μέτρα δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από μένα. Δεν είμαι ακόμα σε θέση να το κάνω. Αλλά όταν εξέταζα το ιστορικό του πώς διαχειριστήκαμε το κοινωτικό κεκτημένο, Ε, ξεπλάγει να δω ότι το θέμα του ύδατος ε, η οδηγία υιοθετήθηκε το 2000 ενώ άλλες οδηγίες ε, για χημικές ουσίες και λοιπά ήταν προηγουμένως και ξεπλάγει ότι η οδηγία ήταν του 2000 μια προσέγγιση πολύ βασική συνολικά συστήματα αξιολόγησης διαμεθοριακή συνεργασία, ένα θέμα που πιστεύω θα εξετάσω προσεκτικά. Προγραμματισμός και διαβούλευσης για το προγραμματισμό. Η αρχή του οριπένων πληρώνει. Επίσης, η επιβολή τιμής για όλα τα αποθέματα ύδατος, σημαντικό επίσης. Ε, επίσης ξεσορρόψει με άλλους τομείς και άλλες πολιτικές. Όλα αυτά είναι τμήμα του σκεπτικού που ακολουθεί η οδηγία αυτή. Η αποτελεσματικότητα λοιπόν όσον αφορά την τιμή δεν έχει εξασθεί επαρκώς. Αλλά σε σχέση με την νομοθεσία που υιοθετήσαμε, που υπάρχει αυτή τη στιγμή, μπορεί να είστε σίγουροι ότι θα εξετάσω πολύ προσεκτικά όλα τα θέματα της εφαρμογής της. Και η πολιτική μου είναι ότι θα πρέπει να είναι απλά για τα κράτη-μέλη, άμεσα, χρήσιμα και προσπαθώ να βοηθήσουμε. Ε, θα πρέπει βέβαια όλα αυτά να τα κάνουμε για προς όφελος όλων και όχι εις βάρος. Αστέως ε, επίτροπος για έρευνα και επιστήμη, για εξηγήστε μου, ποια είναι τα καινοτομικά μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, γεωργία ή και τον οικιστικό τομέα για να μειωθεί ή κατανάλωση ύδατος. Και επίσης η κατασπατάληση του ύδατος. Κατασπαταλούμε πολύ νερό στην Ευρώπη. Το 70% των υδάτων χρησιμοποιούνται από τη Γεωργία στην Ευρώπη. Πώς μπορούν οι νέες τεχνολογίες να εισαχθούν σε συνεργασία με τη Γεωργία, παραδείγματος χάνει και με άλλους τομείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. You are pretty Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό νέες τεχνολογικές εξελίξεις να βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι ενδυναμώνουμε την προσέγγιση μας προς όφελος όλων αυτών που προαναφέρατε. Είναι σημαντικό λοιπόν να πούμε ότι δεν μιλάμε μόνο για βιοτεχνολογία, νανοτεχνολογία, πληροφορική που είναι οι πιο προηγμένες τεχνολογίες. Όχι, πρέπει να ξέρουμε πώς μπορούμε κατά τον δικότερο τρόπο να χρησιμοποιήσουμε νέες τεχνολογικές αποφάσεις στους τομείς που προαναφέρατε. Γεωργία Φερρυπίν. Πάρα πολύ σημαντικό. And τις σας για την αποτελεσματική χρήση των υδάτων. Είναι πραγματικά ένα θέμα που πρέπει να ε, τύχει της προσοχής μας. Αλλά πάλι χρειαζόμαστε μια ολιστική προσέγγιση. Τιμή, μέτρα για τη ζήτηση, τεχνολογικά μέτρα, συμπεριφορά κλπ. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Και προς τα εκεί θα ήθελα να κι εγώ. Ευχαριστώ. Πείτε, Λίζε, για το φινάλε τώρα. Ευχαριστώ. Εξότιμη κύριε υποψήφια επίτροπε, έχω μια ερώτηση σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με το άρθρο 225 της συνθήκης, τέος 152 άρθρο, το Κοινοβούλιο έχει ένα έμεσο δικαίωμα πρωτοβουλίας και στη γραπτή σας απάντηση λέτε «Λαμβάνω υπόψη» Αλλά η συνθήκη λέει κάτι παραπάνω και ξέρετε σίγουρα ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη διαπραγματευτεί το θέμα με τον πρόεδρο της Επιτροπής, κύριο Παρόζο. Και θα θέλαμε καταρχήν, υπάρχουν ξέρετε αλλά καταρχήν όταν υποβάλλουμε μία ε, πρόταση με στασμένη πλειοψηφία να μας υποβάλει σχετικά την πρόταση την νομοθετική κομισιόν. Θα το κάνετε και εσείς συγκεκριμένα και θα υποστηρίξετε ε, το θέμα αυτό πριν από τη πληροφορία για την Κομισιόν το τέλος του μηνός. Ευχαριστώ. Απάντηση. Ε, θεωρώ ότι η συνδείξη της αγώνας είναι ξεκάθαρη. Λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί με πλειοψηφία των μελών του να υποβάλει κάποια κατάλληλα μέτρα που θεωρεί ότι πρέπει να είναι αντικείμενο της δράσης των ευρωπαϊκών ε, κρατών. Και αν δεν υποβάλει σχετική πρόταση Κομισιόν θα πρέπει να ε, αιτιολογήσει προς το Κοινοβούλιο γιατί δεν το κάνει. Διαπραγματευτήκαμε διαμακρών αυτή τη συνθήκη και νομίζω θα πρέπει να την εφαρμόσουμε τώρα. Και προσωπικά εγώ πιστεύω ότι αν η πρόταση του Κοινοβουλίου παρουσιαστεί όπως το είπατε εσείς θα πρέπει να τη λάβουμε πάρα πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Και θυμάμαι ότι η πρώτη Επιτροπή Παρόσο είχε πολύ καλό αποτέλεσμα τελικά όσον αφορά αυτό το θέμα. Κατά βάση Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα μεταξύ μας εδώ, αλλά είναι ένα πρόβλημα θεσμικής συμφωνίας μεταξύ Κοινοβουλίου και Κομισιόν γενικά, μια θεσμική συμφωνία δηλαδή. Α, θεωρώ όμως ότι ο πρόεδρος Μπαρόσο όταν είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ειδική εταιρική σχέση με το Κοινοβούλιο, το θεωρούσε πάρα πολύ σοβαρό. Και ειδική εταιρική σχέση σημαίνει και ανοιχτή συνεργασία. Και αυτό σημαίνει ότι όταν έχει υποβληθεί μια σοβαρή πρόταση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί εξίσου σοβαρά. Ευχαριστώ. Συμπραγματική ερώτηση. Ναι, έχετε δίκιο. Αναφέρεται αυτό στην συνθήκη ότι θα πρέπει η Κομισιόν να αιτιολογήσει γιατί δεν υποβάλλει μια πρόταση. Αλλά θα ήθελα να ξέρω τι θα κάνετε εσείς στον τομέα για τον οποίο θα είστε αρμόδιος, τι θα προτείνετε στο συλλογικό σώμα της Κομισιόν και ποια θα είναι τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήσετε έναντι του κυρίου Μπαρόσα. Για ποιους λόγους δεν θα υποβάλει ε, η Κομισιόν μια πρόταση. Μπορείτε να μας εγγυηθείτε ότι η αιτιολόγηση δεν θα είναι ότι μου τηλεφωνήσαν από το Βερολίνο, από το Λονδίνο, από το Παρίσι και αυτό το κάνω. Δηλαδή να συνεργαστείτε με το Κοινοβούλιο ακόμα και να αντίθετο Συμβούλιο. Ε, μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι οπωσδήποτε ε, το τηλεφώνημα ούτε από το Βερολίνο, από το Λονδίνο, ούτε από τη Λουμπλιάνα θα με αποτρέψει στην λήψη μια απόφαση. Αλλά επαναλαμβάνω αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να ε, αντιμετωπιστεί στις σχέσεις μεταξύ της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου γενικά. Αν έχετε εσείς μια πρόταση που βασίζεται σε πλειοψηφία που είναι πολύ σοβαρή, μπορώ πραγματικά να λάβω τη δέσμευση εδώ. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι θα ακολουθήσω τη συνθήκη που ισχύει. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να σας υποσχεθώ εγώ εδώ, αλλά νομίζω ότι αυτού του τύπου οι προτάσεις θα πρέπει να εξεταστούν πάρα πολύ σοβαρά. Και αν η Κομισιόν πει όχι, Και εδώ θα ήθελα να σας αναφέρω στα αποτελέσματα της πρώτης ε, Επιτροπής Περόσο. Αλλά εάν, λέω, θα πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή αιτιολόγηση. Όλα τα άλλα θα πρέπει να είναι αντικείμενα συμπληρωματικών εμφανισμών μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Πρόεδρο, αγαπητοί συνάδελφοι, βρισκόμαστε στο τέλο του χρόνου τη ερωτήσεων. Σα ευχαριστώ πολύ που καταφέραμε να τηρήσουμε του κανόνε και να μείνουμε και μέσα στα χρονικά όρια που έχουμε που και που κάποιος ε, συνάδελφος έλειψε. Κάνουμε οικονομία λοιπόν τα πέντε του λεπτά. Νομίζω ότι ο υποψήφιο ε, επίτροπος Ποτότσια εργάζεται πάρα πολύ σκληρά Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Από εδώ βλέπω όλα αυτά τα χαρτιά που έγραψε. Μας είπε ότι είναι πράσινο ε, η Ευρωπαϊκή πυρο και ο πλανήτη είναι μπλε, αλλά εδώ πέρα λέω, βλέπω ένα σωρό χρώματα και κίτρινο και μπλε και πράσινο και ροζ και ό,τι θέλετε. And I think we touched in this... Uh, και νομίζω στις τρεις αυτές τις ώρες ε, κάναμε πραγματικά μία, ένα γύρο πολλών θεμάτων που μας απασχολούν και είναι σημαντικά για τις δικές μας θέσεις. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας και ευχαριστώ τον Επίτροπο για τις απαντήσεις σας. Λοιπόν, στο τέλος μας είπατε ότι στα 5 λεπτά θα μας συνεχίσετε την ερώτηση του προσωπικού σας ε, προγράμματος δράση για να σώσετε το περιβάλλον. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η συνήθιση θερμοκρασία στο σαλόνι σας και στο γραφείο σας, γιατί εδώ στην αίθουσα είναι 25 βαθμοί Κελσίου. Αρκετά ζεστά δηλαδή. Λοιπόν, το περιβαλλοντολογικό σύστημα διαχείρισης του περιβάλλον ε, στο κοινοβούλιο θα μπορούσε να βελτιωθεί. Ξέρω ότι οι κυρίες κάπως κρυώνουν πιο εύκολα. Okay, anyway, I stop. I think I give... Εντάξει, εντάξει, δεν θα συνεχίσω. Θα δώσω το λόγο για την τελική παρουσίαση.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 στην αρχή και στο τέλος της συνεδρίας θα έπρεπε να μετρηθεί η θερμοκρασία. Πάντως ε, η θερμοκρασία, κατάλληλη θερμοκρασία εργασίας είναι 21 βαθμοί. Δυστυχώς εγώ είμαι άνθρωπος που προτιμώ θερμότερα κλίματα από ότι τα ψυχρότερα, αλλά προέρχομαι από μια χώρα όπου είμαστε συνηθισμένοι στις χαμηλές θερμοκρασίες. Αν θέλετε όμως θα μπορούσα να σας πω δύο λόγια για το τέλος αυτής της ακρόασης. Όταν ε, διάβασα όλη αυτή την πανοπλία οδηγιών, εγγράφων και νέων ε, συντομεύσεων ακροστοιχείων που πρέπει να συνηθίσω, ε, πριν να ξεκινήσω και να μπω σε περισσότερε λεπτομέρειες και σε πιο οριζόντια έγγραφα, πριν να αρχίσω να μελετώ τα θέματα που συνδέονται με το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο δράση 2007 ε, και το EPR 2008 και κάποια από τα έγγραφα κτλ. Ε, ε Είπαμε, είπα ως προτεραιότητες εγώ από μόνος μου ότι θα έπρεπε να είναι πιο σημαντικά στην ατζέντα τα θέματα περιβάλλοντος. Η βιωσιμότητα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ολιστικά και οριζόντιες πολιτικές θα πρέπει να γίνονται σε συνεργασία με τις κλιματικές αλλαγές και με όλες τις άλλες πολιτικές. Όπως σας είπα, εγώ βασικά έχω να κάνω με θέματα παγορημέτρα, παγορευτικά, ενώ οι άλλοι έχουν κίνητρα στα χέρια τους που εγώ θα θέλω να συνδυάσουμε. Ζούμε σε μια οικονομία της αγοράς και βέβαια θα πρέπει να δίνονται πάντοτε ευκαιρίες απασχόλησης. Το περιβάλλον θα πρέπει να συμβαδίζει με την οικονομία και όχι να είναι εναντίον τη. Το πρόγραμμα της Οικονομία χωρίς άνθρακα θα πρέπει να οδηγήσει σε μια οικονομία που θα είναι ε, ε, ε, επαρκής όσον αφορά τους πόρους και την ενέργεια. Θα πρέ... Είναι σημαντικό να αυξηθεί η άμεση χρηματοδότηση για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά είναι πιο σημαντικό όλα τα χρηματοδοτικά μέσα να χρησιμοποιούνται με τρόπο συνεπή με την ε, προσέγγιση βιωσιμότητας και τους περιβαλλοντικούς στόχους. Πιο ενεργή διεθνή συμμετοχή θα πρέπει να υπάρξει, γιατί πολλά ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο σφαιρικά και ούτω καθεξής. Και τα υπόλοιπα αφορούν πιο συγκεκριμένα στοιχεία για, κάθε, για το χαρτοφυλάκιο και ε, πραγματικά προσέβλεπα στη σημερινή μας συζήτηση γιατί ελπίζω πως θα είναι η αρχή για μια καλή συνεργασία κατά τη διάρκεια των επομένων πέντε ετών. Ειλικρινά πιστεύω πως θα μπορούσε κάτι τέτοιο να γίνει. Όπως σας είπα θα είμαι πάντα ανοιχτός σε οποιαδήποτε πρόταση και οποιαδήποτε πρόσκληση να έρθω να σας επισκεφτώ και να συζητήσουμε τα θέματα. Ε, και αν θέλετε τέλος Τελικά να σας πω την ιστορία του Πράιος. Ο γιος μου, 13 Νοεμβρίου, 13 η ώρα. Και σήμερα είναι 13, 13 ε, του Ιανουαρίου, 13 η ώρα ήταν η ακρόαση. Ο γιος μου τράκαρε εκείνη την ημέρα και εγώ σήμερα είχα ακρόαση. Ε, είπα λοιπόν και σκέφτηκα άμα ήταν κακό το κάρμα έπρεπε να το σπάσω σήμερα. Και σας ευχαριστώ για όλα σήμερα. Ελπίζω πραγματικά να έχουμε καλή συνεργασία για τα επόμενα ε, χρόνια. Thank Σας ευχαριστώ συνάδελφοι, ευχαριστούμε υποψήφια Επίτροπε Ποτότνικ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι τρεις ώρες που περάσαμε μαζί. Τέλος της ακρόσης και καλό τους συντονιστές να, να συναντηθούν σε μισή ώρα στην 1G2 για την αξιολόγηση της ακρόσης. Ευχαριστώ.